Λοιπόν, συνάδελφοι, αν έχετε την καλοσύνη να καθίσετε για να ξεκινήσουμε. Δεν έχουν έρθει ακόμα οι υπουργοί. Ε, παρ' όλα αυτά όμως θα ξεκινήσουμε με τις ε, ανακοινώσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Και θα αναφερθώ τώρα στο γλωσσικό καθεστώς, ε, γαλλικά, εστονικά, ε, λετονικά, μαλτέζικα, κροατικά και γκέλικ δεν υπάρχουν σήμερα. Αλλά θέλω να σας πω επίσης ότι με βάση μια επιστολή που ίσως και να έχετε διαβάσει μερικοί από εσά και μετά από συζητήσεις ε, που έγιναν σε επίπεδο συντονιστών, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα Έχουμε πολλή δουλειά. Σήμερα ξεκινάμε στις 2.30 ε, για να βολέψουμε κάπως τη συνάντησή μας και τον Βέλγο Υπουργό και έχουμε και την Πέμπτη τα απόγευμα ε, συνάντηση τελείως απρόβλεπτα, άρα δηλαδή τέσσερις ε, συναντήσεις επιτροπής το Μάιο και θα έχουμε και άλλη μία συνάντηση στο Στρασβούργο. Και ίσως λοιπόν έχετε ήδη δει ότι είχαμε πέντε συνεδριάσεις επιτροπής μας τον Απρίλιο και ο λόγος που τα λέω όλα αυτά είναι ότι ε, κάθε εβδομάδα μας κατατίθενται 5-10 εβδομάδες από την Επιτροπή και θέλω να σας ε, διαβεβαιώσω ότι δεν είναι ότι ε, πολλαπλασιάζουμε τις συναντήσεις χωρίς λόγο, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε το νομοθετικό φόρτο. Και προσπαθούμε να ανταποκριτούμε όσο καλύτερα μπορούμε και στις διάφορες προτάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, όπως και κάνουμε σήμερα. Αυτά ήθελα να σας πω. Τώρα αν έχετε κάποια ερώτηση, κάποια ε, προτίμηση, ε, παρακαλώ να μην ε, διστάσετε να με το πείτε, ακόμα και αν δεν ελέγχετε στις συνεδρίες των συντονιστών. Λοιπόν, άλλα θέματα που θέλω να φέρω πολύ γρήγορα. Έχουμε ε, μια, ένα τηλεοπτικό κανάλι από τη Γεωργία που ε, θέλει να γυρίσει κάπως ε, κάποιες σκηνές από τις ενδρίασή μας, κυρίως για το τελευταίο κομμάτι της ημερησίας διάταξης. Επίσης, ο Τζόλ Μπεργκερών... από την ομάδα FTT έχει οριστεί εισηγητής για την έκθεση πρωτοβουλίας για τα συστήματα εγκλισμού και τις προϋποθέσεις. Η Κριστή Ρεβόντολό έχει οριστεί εισηγήτρια για την ενδιάμεση έκθεση πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υγεία κατά των γυναικών και την εσωτερική και κατοίκον βία. Ο κύριος Αγγιλάρ έχει οριστεί ο ε, συντάκτης της γνωμοδότησης προς την κατεύθυνση του καθεστώτος, του οριστικού καθεστώτους ε, ΦΠΑ και αντιμετώπιση απατών με το ΦΠΑ. Κυρίες και κύριοι, Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορέσαμε να ε, προσκαλέσουμε και η πρόσκλησή μας έγινε αποδεκτή από τους δύο Βέλγους υπουργούς ε, και αυτό μετά τις ε, πρόσφατες ολέκτριες τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρες στις Βρυξέλλες το Μάρτιο στις 22 Μαρτίου. Θα έχουμε συζήτηση με τον κύριο Ζαμπόν, αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό εσωτερικών και τον κύριο Κρουν τον Βέλγο υπουργό δικαιοσύνης. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τους ε, δυο σας, ελπίζω να πρόφερα και καλά τα ονόματά σας. Αγαπητοί συνάλφοι, όπως είπα, έχουμε σοκαριστεί όλοι από, τις, ε, από τα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα πρόσφατα. Η δική μας Επιτροπή ε, θεώρησε ότι σε θεσμικό επίπεδο έπρεπε να απευθυνθεί στους δύο υπουργού. Και εμείς θέλουμε να ενημερωθούμε γενικότερα για το ρόλο του Συμβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Θελήσαμε επίσης να συζητήσουμε με τους υπουργούς, να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί τυχαίνει να βρίσκεται μεταξύ άλλων και η έδρα του δικού μας του Κοινοβουλίου εδώ. Και θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς διαδραματίζεται. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και οι δυο σα και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, γιατί δεν έχουμε και άπλετο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα μου επιτρέπετε να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Ζαμπό, ο οποίος είναι η αναπληρωτής Πρωθυπουργό και Υπουργό Ασφάλειας και Ιστορικών Υποθέσεων. Θα μιλήσει περίπου για 6 λεπτά και μετά θα έχουμε ερωταπαντήσεις. Ε, αγαπητέ Ζαν, σε ευχαριστούμε που ήρθατε και χαίρομαστε πάρα πολύ και ευχαριστούμε για όλα αυτά που συνέβησαν μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλωσορίζω και όλους σας. Ε, θέλω να σας πω ότι είναι τιμή για μένα το ότι μπορώ να βρίσκομαι σήμερα το απόγευμα εδώ κάτω από αυτές τις ε, τραγικές συνθήκες. Θα μιλήσω στα αγγλικά, εισαγωγικά, προφανώς και μπορώ να χρησιμοποιήσω την ε, μητρική μου γλώσσα που είναι το και αν θέλετε μπορείτε να γυρίσετε εσείς ε, στην ε, δική σας τη μητρική γλώσσα. Έχουν περάσει περίπου δύο μήνες από τότε που οι δύο τρομοκράτες επιτέθηκαν πρώτα στο αεροδρόμιο του Ζάβεντεμ και μετά στο σταθμό του μετρό στο Μάλμπεκ κοντά στο Κοινοβούλιο. Τρενήσαμε πάρα πολλά θύματα, 32 νεκροί, εκατοντάδε τραυματίες από πολλά κράτη συμπεριλαμβανομένων και ανθρώπων που εργάζονται για τους ε, ε, νοσιακούς θεσμούς. Πάρα πολλοί τραυματίες, ακόμα και σήμερα βρίσκονται στην εντατική και πολλά από τα θύματα, από τους τραυματίες, ε, τραυματίστηκαν διαβίου από αυτή την δειλή επίθεση, από την επίθεση κατά των αξιών της ανοιχτής ε, δημοκρατικής ε, κοινωνίας, την οποία εμείς υπερασπιζόμαστε. Ήταν λοιπόν η χειρότερη τρομοκρατική επίθεση που έλαβε ποτέ χώρα στη χώρα μας ήταν το δικό μας, η δική μας 11η Σεπτεμβρίου Είχαμε τρεις ε, ημέρες εθνικού πέντους και θα ήθελα στο όνομα της ε, βελγικής κυβέρνησης και των Ευρωπαίων εταίρων μας, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών θεσμών, να σας ευχαριστήσω όλους ε, για την αλληλεγγύη που επιδείξατε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα συλληπιτήρια που εκφράσατε προς το βελγικό λαό. Πέρα λοιπόν από τον ανθρώπινο πόνο ε, προκλήθηκαν και πολλές υλικέ ζημιές. Το αεροδρόμιο του Ζαβεντέ αναγκαστικά έκλεισε για κάποιο χρονικό διάστημα και έκλεισαν επίσης και κάποιες γραμμές του μετρό. Την ίδια την ημέρα της επίθεσης η βελγική κυβέρνηση στο βαθμό του δυνατού προτίμησε να μην προκαλέσει φόβο γιατί ακριβώς αυτό ήθελαν να εμπνεύσουν οι τρομοκράτες. Ε, δηλαδή δεν παρέλυσαν οι Βρυξέλλες, του αντίον οργανώσαμε τις δημόσιες μεταφορές ε, με ελεγχόμενο τρόπο, με επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Τώρα το μετρό και το αεροδρόμιο έχουν αρχίσει πάλι να λειτουργούν. Το μετρό λειτουργεί πλήρως. Άνοιξε και πάλι ο σταθμός του Μάλμπεκ. Το αεροδρόμιο απ' την άλλη ε, δεν έχει επανέλθει πλήρως, αλλά θα επανέλθουμε πλήρως. Αμέσως μετά τις επιθέσεις ε, ανακοινώσαμε ύψιστο βαθμό συναγερμού για το σύνολο της χώρας. Τώρα, μετά από ένα μήνα, είμαστε στο, στην βαθμίδα υπαριθμών 3. Είναι το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που ερμηνεύεται ως ε, σοβαρή απειλή με ενδεχόμενο επίθεσης αλλά χωρίς να γνωρίζουμε πού και πότε μπορεί να λάβει η χώρα η επίθεση αυτή. Οι έρευνες που και ποτε μπορει να λαβει χωρα η μετά τις επιθέσεις συνεχίζονται πλήρως και θα ήθελα να σας πω ότι δουλεύουμε ολόκληρο το 24ωρο για τα θέματα αυτά. Έχουμε προβεί σε επιδρομές, σε συλλήψεις υπόπτων και ευχαριστούμε την κοινή κυβερνητική ομάδα η οποία συναισθήθη αμέσω μετά τι επιθέσει. Αναφέρομαι στην ομάδα ε, την κοινή από βελγικέ και γαλλικέ αρχέ. Αποδείχθηκε ότι αυτή η τρομοκρατική ομάδα ήθελε να ξαναεπιτεθεί στη Γαλλία αλλά χάρη στην ταχύτατη επέμβαση των δυνάμεων ασφαλεία μπορέσαμε να προλάβουμε κάτι τέτοιο και γι' αυτό το λόγο αυτοί οι τρομοκράτες, ανταυτού δηλαδή, ε, προτίμησαν να επιτεθούν στις Βρυξέλλες. Η συνεχιζόμενη απειλή σημαίνει ότι ορισμένες στρατηγικής σημασίες περιοχές εξακολουθούν να είναι υποστενή παρακολούθηση. Αναφέρομαι στους πυρηνικούς σταθμούς, στο αεροδρόμιο, ε, στις δημόσιες μεταφορές υπάρχουν και ήπιοι στόχοι όπως είναι οι κινηματογράφοι και αυτοί ελέγχονται πιο στενά. Επίσης, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραμένει και να επικρατεί ασφάλεια σε ολόκληρη τη χώρα. Ε, πριν από τις επιθέσεις Βρυξέλλες, ε, εδώ ελήφθη μια ολόκληρη σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα 30 αριθμούν τα μέτρα αυτά. 12 ανακοινώθηκαν στις αρχές ε, του 2015 μετά την επίδυση στο Παρίσι και 18 επιπρόσθετα μέτρα ακολούθησαν μετά την επίθεση του Νοεμβρίου. Ε, το 2015 μιλάμε για 200 εκατομμύρια που διατέθηκαν και το 2016 το ποσό αυτό ανέρχεται πλέον σε 400 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διατίθενται για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ε, κάποια από αυτά τα κονδύλια δόθηκαν φάπαξ ε, και άλλα θα έχουν μια χρονική διάρκεια γιατί ε, εκταμιεύονται για έργα υποδομής. Οι αποφάσεις που έλαβε η βελγική κυβέρνηση ήταν η εξή. Ο Υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων μπορεί να αποσύρει ταυτότητες αν δηλαδή θέλει κάποιο να πάει στη Συρία, είναι ύποπτο μάλλον ότι μπορεί να μεταβεί στη Συρία, μπορούμε να το αποσύρουμε την ταυτότητά του, το διαβατήριό του. Η, μάλλον, εμείς την ταυτότητα, το διαβατήριο μπορούν να το ε, πράξουν οι συνάδελφοί μας αν υπάρχει κίνδυνο, σας είπα, και υπάρχει υποψία. Εξάλλου, ανανεώθηκε το πρόγραμμα για την ρίζοσπαστικοποίηση, αναπτύχθηκαν δυνάμεις του στρατού, ενισχύθηκαν οι αστυνομικοί έλεγχοι στα σύνορα και το συντομότερο δυνατόν ε, θα θεσπίσουμε και στο Βέλγιο το νόμο περί μητρώου επιβατών για το PNR. Στο μέλλον θα λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη μας ε, μέτρα που έχουν σχέση με τις ε, προπληρωμένες κάρτες ε, τηλεφώνου, τις ανώνυμες, μάλλον αυτές δεν θα μπορεί κανείς πλέον να τις αγοράζει. Μετά το Παρίσι είχαμε πάρα πολλές ε, ενδείξεις ότι η περιοχή του Μόλεμπεκ ήταν προβληματική, αλλά θέλω να σας πω ότι εμείς δεν ασχοληθήκαμε μόνο με το Μόλεμπεκ, ασχοληθήκαμε και με άλλα 7 άλλες 7 ε, περιοχές ε, στο κανάλι, παράλληλα στο κανάλι των Βρυξελών. Το Βέλγιο ε, μάχεται κατά το ISIS με σκάφη και με στρατιωτικά αεροπλάνα. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυξημένο επίπεδο ασφάλειας στη χώρα μας. Κυρίε και κύριοι, οι τρομοκράτες επιθυμούν να επιφέρουν διαίρεση και δεν πρέπει να πέσουμε μέσα σε αυτή την παγίδα. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση που διεξάγεται δημόσια είναι πάρα πολύ σκληρή. Έχει ασκηθεί σκληρή κριτική στο Βέλγιο. Εγώ ως υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων θέλησα να σας διαβεβαιώσω ότι στο Βέλγιο όλες οι υπηρεσίες συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα ε, κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες. Αυτό το θέμα, το φαινόμενο των ε, ξένων μαχητών, ε, των foreign fighters είναι πολύ ε, δύσκολο να αντιμετωπιστεί και το θέμα δεν είναι μόνο η ρίζοσπαστικοποίηση των ανθρώπων αυτών, δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν ε, κλειστέ κοινωνίε μέσα στην ευρύτερη κοινωνία. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε και τι μετακινήσει των ανθρώπων αυτών. Θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στι υπηρεσίε μυστικές υπηρεσίες να παρακολουθούνται και οι άνθρωποι που επιστρέφουν από την Συρία. Θα πρέπει να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις παράνομες ε, χρηματοδοτήσεις. Ε, για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τρίτες χώρες. Όλα αυτά λοιπόν είναι καθοριστική σημασία για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η τρομοκρατία. Η λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε δεν είναι απλή, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και εμεί θέλουμε να διαθέσουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Φοβάμαι ότι η κοινωνία θα κληθεί ε, να πληρώσει στο μέλλον μεγαλύτερο τίμημα για την ασφάλεια από αυτό που καταβάλει τώρα. Ασκείται βέβαια έντονη κριτική για το τι έκαναν οι βελγικές αρχές. Η κριτική αυτή εκφράζεται στα μέσα ενημέρωσης και εντός και εκτός Βελγίου. Η κριτική συνεχίζεται και ορισμένα πράγματα αναμφίβολα μπορούν να βελτιωθούν. Γνωρίζετε ότι στο Βελγικό Κοινοβούλιο συναισθήθη μια επιτροπή για να εξετάσει όλες τις πτυχές ε, της επίθεσης. Στο ίδιο το Βέλγιο ε, θα αναζητήσουμε και θα ψάξουμε τη δική μας ε, την επίδοση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την, τις ελλείψεις μας να έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Όσον αφορά στην Ευρώπη και όσον αφορά αυτά που γνωρίζουμε τώρα για τους τρομοκράτες και τις μετακινήσεις τους, είναι σαφές ότι η τρομοκρατία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο εφόσον υπάρχει συνεργασία τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ε, το Φεβρουάριο του 2015 στο Συμβούλιο ε, που συνεκλήθη αμέσως μετά την επίθεση στο Παρίσι, εκεί ελήφθησαν μέτρα τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Έχουν καταρτιστεί μία σειρά καταλόγων, μεταξύ αυτών προβλέπεται η ταχύτατη, η μη καθυστερημένη θέσπιση της οδηγίας περί Μητρόπιβατών. Επίσης, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, ανταλλαγή πληροφοριών και σε επίπεδο Europol, λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας ε, των τρομοκρατών και για την παρουσίαση ενός διαφορετικού αφηγήματος. Όπως ε, ξέρετε, όσον αφορά στην ασφάλεια, εμείς ε, έχουμε την προεδρία των G11 και των G11 και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε την ε, τρομοκρατία. Τώρα, θα ήθελα να πω και ορισμένε λεπτομέρειε. Δηλαδή, είμαι ιδιαίτερα ευτυχή που η οδηγία επιβατών μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς επιτέλους ε, αυτή η οδηγία εγκρίθηκε στις 14 Απριλίου με συντριπτική πλειοψηφία. Τώρα το Μητρό Επιβατών δεν είναι αναμφίβολα η μαγική λύση, αλλά είναι εν πάση περιπτώσει μια λύση που θα βοηθήσει τις αρχές ασφαλείας να συγκεντρώνουν από κοινού και να αναλύουν από κοινού τα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται και με άλλες πηγές δεδομένων και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εξάλλου, το Βέλγιο επιθυμεί να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η οδηγία αυτή να επιτρέπει να χρησιμοποιούνται δεδομένα και μέσα από τις εσωτερικές πτήσεις ε, στην Ευρώπη. Είμαστε στην τελευταία φάση της ψηφιακής επεξεργασίας. Όσον αφορά στα σύνορα, οι Ευρωπαίοι ε, πολίτες τα ελέγχονται στα εξωτερικά σύνορα με βάση όμως κάποιους δείκτες κινδύνου. Αποφασίστηκε στο ε, Συμβούλιο ε, το που έλαβε χώρα στις 24 Τρίτου αποφασίσαμε να εξετάζουμε συστηματικά κατά πόσον ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν απειλή. Οι νέοι κανόνες θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο αυτή η νέα νομοθεσία να τεθεί ε, σε ισχύ πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές για να αρχίσουμε να την ε, εφαρμόζουμε το συντομότερο δυνατόν λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας της κατάστασης, οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα ήταν ανεύθυνη. Η ανταλλαγή πληροφοριών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι κάτι που θέλω να θίξω. Ο συντονιστής ε, John Παντεκέκοβερ, συντονιστής για θέματα τρομοκρατίας, είπε την προηγούμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο ότι ακόμα δεν χρησιμοποιούνται πλήρω τα ευρωπαϊκά εργαλεία όπω είναι ε, το σύστημα ε, πληροφοριών του Schengen και η Europol. τι τελευταίε εβδομάδε. είδαμε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με το Κέντρο αντιτρομοκρατία της Europol. Στι αρχές αυτού του μήνα το Βέλγιο σε συνεργασία με τη Europol οργάνωσαν μια επιχειρησιακή συνάντηση εμπειρογνωμόνων τρομοκρατία από τα κράτη-μέλη ε, συνάντηση αυτών με εμπειρογνώμονες της Europol για να ανταλλάξουν πληροφορίες. Εξάλλου, το Βέλγιο ανέκαθεν πίεζε για μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και για πάρα πολλά χρόνια ήταν μία από τις χώρες οι οποίες έδεκε τις περισσότερες πληροφορίες στη Europol. Η εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει μας πείθει ότι πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μετά από τις επιθέσεις του Νοεμβρίου στο Παρίσι μάθαμε κάτι πολύ χρήσιμο που αφορά στη χρήση του συστήματος πληροφοριών του Schengen και τα γραφεία Sirene στο πλαίσιο της ε, της αντιμετώπισης των ξένων μαχητών. Έχουμε εντοπίσει ορισμένα σημαντικά θέματα για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα SIS, το SIS. Τώρα πλέον ε, είμαστε σίγουροι ότι το σύστημα αυτό πρέπει να εφαρμοστεί από το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. Εξάλλου, πρέπει να υπάρχει καλύτερη συμβατότητα ανάμεσα ε, στις τράπεζες δεδομένων. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από το Συμβούλιο ε, Δικαιοσύνης και Ασφάλειας την προηγούμενη εβδομάδα ε, συμφώνησε ότι θα πρέπει ε, να υπάρχουν καλύτερα συστήματα πληροφοριών, να είναι περισσότερο συμβατά μεταξύ τους, γιατί πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα ε, κατά τις επόμενες εβδομάδες, το επόμενο Συμβούλιο του Ιουλίου, αλλά και σε συναντήσεις ε, εμπειρογνωμόνων. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε ε, σημαντικές αποφάσεις για τα το ποια είναι τα σημεία αυτά που αφορούν στην αποκαλούμενη διαλειτουργικότητα, στο κατά πόσο δηλαδή είναι συμβατά τα συστήματα μεταξύ τους. Όσον αφορά στο διαδίκτυο, η Europol έχει συστήσει ένα πλαίσιο, έχει δουλέψει πολύ σκληρά γι' αυτό και ε, το φόρουμ πληροφορικής προσβλέπω ότι θα προσφέρει και αυτό πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σχεδόν σε όλες τις έρευνε που κάναμε για την τρομοκρατία είδαμε το διαδίκτυο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, η συνεργασία ανάμεσα στι κυβερνήσει, αλλά και τους παρόχους ε, του διαδικτύου, αυτό είναι απολύτω απαραίτητο. Και δεν πρέπει να ε, βλέπουμε μόνο το τι συμβαίνει σε επίπεδο επικοινωνίας ε, και πώς μπορούμε να απομακρύνουμε κακές πληροφορίες από το διαδίκτυο. Αυτό που σας είπα είναι σημαντικό είναι το πώς μπορούμε και εμείς να παρουσιάσουμε το δικό μας το αφήγημα. Το ESCED, η ομάδα αυτή που συστήθηκε στις, ε, το 2015, είναι ένα παράδειγμα αυτού του αφηγήματος. Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο το οποίο στηρίζει το Βέλγιο και με την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε συστήσει ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων για να προσφέρουμε υπηρεσίες, να προσφέρουμε συμβουλές στα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή Επιθυμούμε επίσης ε, να διαπιστώσουμε το πώς μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία στο διαδίκτυο και με τις διάφορες χώρες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Κυρίε και κύριοι, έχουν γίνει πάρα πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπολείπονται όμως ακόμα πολλά. Εγώ σας ανέφερα κάποιους από τους τομείς ε, στους οποίους δραστηριοποιούμεθα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό, εφόσον βρισκόμαστε στο Βέλγιο, να μην περιζόμαστε σε λόγια, αλλά να περάσουμε στις πράξεις. Ας ε, δραστηριοποιηθούμε για να έχουμε γρήγορη επιτυχία και πιστεύω ότι αυτό το περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να γίνει ανταλλαγή απόψεων βεβαίω και πάρα πολλά είναι τα μέλη που θέλουν να μιλήσουν. Ο κύριο Χέιν θα πάρει τώρα το λόγο για 10-15 λεπτά. Σίγουρα θα υπάρξουν πολλέ απαντήσει στα μέλη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά τη Μαδρίτη, το Λονδίνο και το Παρίσι, τρομοκράτες στις Βρυξέλλες, στην πρωτεύουσά σας, στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βελγική κυβέρνηση έχει πλήρη συνέστηση αυτής της διάστασης. Το αεροδρόμιο και ο σταθμός του μετρό Μάλμπεκ είναι χώροι που χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέλη των δικών θεσμικών οργάνων, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που ανήκουν σε όλους μας. Βεβαίως η ευρωπαϊκή διάσταση είναι η μία πτυχή της υπόθεσης ε, της τρομοκρατικής επίθεσης πριν από ένα μήνα. Τα πρώτα βήματα είναι οι καθημερινοί πολίτες που έχασαν τη, ζωή τους, οι απλοί πολίτες σε αυτούς τους βομβαρδισμούς. Πρόκειται για απειλή στο σύνολο του πληθυσμού, στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο και στην Ευρώπη. Πρέπει να εργαστούμε σε, πάνω σε διάφορα μέτρα και αυτά θα αναπτύξω στα 15 λεπτά που μου έχουν δοθεί. Λίγα σχόλια να κάνω για τις έρευνες και τα προκαταρκτικά συμπεράσματα ως προς τα δίκτυα των τρομοκρατών. Από τον Νοέμβριο του 2015 και τις επιθέσεις στο Παρίσι, όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφοριών στην Ευρώπη εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στα δίκτυα πίσω από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών ήταν ανέκαθεν έντονη και έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο έκτοτε και θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να υπογραμμίσω την εξαιρετική σχέση που έχουμε με τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες, με τις γαλλικές δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Έχουμε κοινέ ερευνητικές ομάδες μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου και έχουμε ε, δουλέψει νυχθημερών μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι. Από τη στιγμή που η δικαστική έρευνα εξελίσσεται, δεν δίναμε να μπω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή για την ανάκριση. Ούτε μπορώ να μιλήσω για τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν. Είναι πολύ νωρί σε σχέση με την ανακριτική διαδικασία. Μπορώ όμως να μοιραστώ ε, ορισμένες παρατηρήσεις. Μετά το Βερβιέ το 2015 το ΝΤΑΕΣ έδειξε τι μπορεί να κάνει. Να δώσει εντολές από τη δική του βάση στη Συρία, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις χώρες στόχου, για να ε, ε, στόχος οι επιθέσεις, οι επιθέσεις στο Παρίσι αλλά και στις Βρυξέλλες παρουσιάσουν διάφορες ομοιότητες, κυρίως λόγω του αριθμού των ατόμων που ασχολήθηκαν ε, με την προετοιμασία, οργάνωση και διάπραξη αυτών των επιθέσεων. Οι παρατηρήσει μας λοιπόν είναι οι εξή. Τρομοκράτε στη Γαλλία και στο Βέλγιο μπήκαν στην ευρωπαϊκή επικράτεια χωρί να τους πιάσουν τα, τα ραντάρ μα, μάλλον χρησιμοποιώντα πλαστά έγγραφα και έχουν εμπειρία από τα σύριακά πεδία μάχη, ε, έγινε σύναψη σχέσεων μεταξύ Γάλλων και Βέλγων τζιχαντιστών που συγκρότησαν γαλλόφωνες ή και φλαμανδόφωνες μεραρχίες, τάγματα να το πω έτσι. Εμπνεύστηκαν από τις επιθέσεις στο Παρίσι για να διαπράξουν τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Έχουμε ήπιους στόχους με στόχο να σκοτώσουν όσο να περισσότερους απλούς πολίτες με ε, εκρηκτικούς μηχανικούς, μηχανισμούς ε, αυτό, ε, ε, που είχαν φτιάξει οι ίδιοι. Όλα αυτά τα σχέδια βέβαια άλλαξαν με τη σύλληψη του Σαλάμ Απντεσλάμ και αναγκάστηκαν οι τρομοκράτες να πάνε στη ε, β' σχέδιο και να χρησιμοποιήσουν τα εκρηκτικά που ήδη είχαν στην κατοχή τους για τις επιθέσεις στις Βρυξάλλες στις Βρυξέλλες. Το προφίλ ε, των ε, επιτιθέμενων έχει διαφορές. Τρία όμως είναι τα σημαντικά στοιχεία. Έχουμε αυτούς που μόλις τελειώνουν το σχολείο, πάνε στη Συρία, ριζοσπαστικοποιούνται και επιστρέφουν περισσότερο ριζοσπαστικοποιημένοι παρά ποτέ. Αυτό είναι το ένα προφίλ. Το δεύτερο προφίλ είναι κάποιοι που δεν τους ξέρουμε, δεν έχουμε ακούσει ποτέ για αυτούς και έχουν διάφορες ταυτότητες. Και το τρίτο προφίλ είναι οι άνθρωποι που έχουν βγει από τις βελγικές φυλακές και πάρα πολύ γρήγορα ριζοσπαστικοποιούνται οι επιθέσεις σε υλικές ε, ε, υποδομές έχουν αυξηθεί από τότε που οι βελγικές υπηρεσίες εντόπισαν ε, το φαινόμενο το 2012. Πολλά μέτρα έχουν ληφθεί έκτοτε για να μειωθεί η ροή των αναχωρήσεων, για να παρακολουθούνται όσοι επιστρέφουν. Στενά, τους τελευταίους μήνες έχει διαμορφωθεί η εικόνα Και έχουμε μια ανεπαρκή αντίδραση του Βελγίου στην, ε, τα, στις τάσεις που διαφαίνονται. Είναι μια εικόνα που πλήττει την, το, τη χώρα, αλλά ε, αδικεί και τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει. Υπάρχει αυτή η εικόνα. Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έγινε κανένα λάθος. Είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε ότι έχουν ληφθεί ε, μέτρα το ένα μετά το άλλο σε όλα τα επίπεδα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι το Βέλγιο παραγνώρισε το θέμα των ξένων ε, τρομοκρατών μαχητών. Οι Βέλγοι υπουργοί, οι βελγικές υπηρεσίες ήταν οι πρώτες που σήμαναν το συναγερμό μεταξύ των ομολόγων τους σε ευρωπαϊκή επικράτεια. Το Βέλγιο ήταν μία από τις πρώτες χώρες που έκανε σαφή αξιολόγηση και είχε σαφή στατιστικά στοιχεία και ζήτησε ριζοσπαστικές αλλαγές στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών μελών. Πολλά θα ήθελα να προσθέσω στην εικόνα που παρουσίασε ο συνάδελφος Υπουργό Εσωτερικών. Η δουλειά των ερευνητών και των εισαγγελικών αρχών έχει καταλήξει σε πολύ ε, καλά αποτελέσματα και φαίνεται αυτό στο διεθνή τύπο. Ο ε, μέσο όρο αριθμός ε, καταδικών για τρομοκρατία ήταν 7 με 8 το χρόνο παλιά που δεν ήταν και λίγο το 2014 όμως κατά, μέσα, ο, κατά μέσο όρο έχουμε 55 καταδίκες για τρομοκρατία. 150 άνθρωποι καταδικάστηκαν το 2015 από τα βελγικά δικαστήρια. Είναι εξαιρετικά υψηλός ο αριθμός αυτός με απόλυτους όρους και είναι πραγματικά ε, εκπληκτικός λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του βελγικού πληθυσμού. Φαίνεται πόσο μεγάλη προτεραιότητα δίνει το Βέλγιο σε όλο αυτό το θέμα. Η βελγική αστυνομία και οι βελγικές εισαγγελικέ και δικαστικές αρχές. Πολλέ αλλαγές έχουν γίνει στην νομοθεσία στο Βέλγιο. Έχει παραταθεί η περίοδος προσωποκράτηση πριν εμφανιστεί ο κατηγορούμενος, ο ύποπτο ενώπιον δικαστού. Μπορεί να υπάρξουν... Ε, έφοδοι της αστυνομίας με εισαγγελέα σε σπίτια και να γίνουν έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ακόμα. Έχουν ε, βελτιωθεί οι τεχνικές διερεύνησης, ανάκρισης, έχει διευρυθεί το πεδίο εφαρμογής των ποινικών αδικημάτων και περιλαμβάνονται εκεί πολύ περισσότερα από ό,τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Έχουμε νέους κανόνες για τη διατήρηση των δεδομένων, σεβόμενοι πάντοτε τις αποφάσεις περί προσωπικών δεδομένων και έχουμε αλλαγές στην νομοθεσία για τις προπληρωμένες κάρτες ε, κινητής τηλεφωνίας. Έχουν γίνει λοιπόν πάρα πολλά βήματα και έχει εξεταστεί και βημακρόν το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης μέσα στη φυλακή. Εφαρμόζεται σχέδιο δράσης, κατάρτιση του προσωφρονιστικού προσωπικού των φυλακών. Έχουμε, θα έχουμε ειδικά τμήματα μέσα στις φυλακές ε, για του ε, καταδίκους για τους οποίους υπάρχει επικίνδυνος να ριζοσπαστικοποιήσουν άλλους ε, ε συγκαταδίκους τους και συγκρατούμενούς τους. Έχουμε καλύτερο εξοπλισμό, καλύτερη νομοθεσία, καλύτερε ερευνητικέ και ανακριτικές ε, τεχνικέ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, μιλούμε ε, για χαρτοφυλάκια που έχουν να κάνουν με την απασχόληση, με τι κοινωνικέ υποθέσει, όλα αυτά που είναι αρμοδιότητα τη τοπική αυτοδιοίκηση ή τη περιφερειακή αυτοδιοίκηση και όχι τη κεντρική κυβέρνηση. Δεν θέλω η της περιφερειακης αυτοδιοικηση και οχι τη κεντρικη κυβερνηση δεν θελω η επιτροπη σα να νομίζει ότι επειδή μα ενδιαφέρει ασφάλεια ασφάλεια και δικαιοσύνη, ασχολούμαστε μόνο με αυτά και δεν ασχολούμαστε με τα λοιπά που μπορεί να σχετίζονται με τη ριζοσπαστικοποίηση. Έχουμε ως χώρα την ισχυρότερη αντίδραση έναντι των ξένων μαχητών από το 2014-2015 και μετά. Στηρίζω τις εργασίες, στηρίζουμε τις εργασίες για τη νέα οδηγία για τα τρομοκρατικά αδικήματα και εμείς έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι προβλέπει αυτή η οδηγία. Θέλουμε ανταλλαγή καλόπρακτικών πρακτικό για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές. Θέλουμε να επεκτείνουμε το ΕΚΡΙΣ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα ποινικά μητρώα, να περιλαμβάνονται εκεί και υπηκόοι τρίτων χωρών και θέλουμε καλύτερη νομοθεσία για την απόκτηση και διάθεση πυροβόλων όπλων την νόμιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν καλύτερη συνεργασία για συγκεκριμένες δικαστικές έρευνες. Η αντιτρομοκρατική μας ε, δράση θα εξαρτάται από στοιχεία που θα έχουν συλλεγεί ηλεκτρονικά για την πρόληψη των επιθέσεων. Αυτό θα συμβαίνει όλο και περισσότερο. Έχουμε την μου στον εθνικό πάροχο υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας και έχουμε σαφείς ε, ε, έχουμε αλλάξει την νομοθεσία σε σχέση με την πρόξιμου και όλου τους παρόχους που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτε. Μόλις την αλλάξαμε, εγκατέλειψαν την κλασική κινητή τηλεφωνία οι τρομοκράτε, και ασχολήθηκαν και άρχισαν να επικοινωνούν με διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικές όπως το Viber για παράδειγμα. Ε, θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις αυτές και να γίνονται σωστές έρευνες με βάση δικαστικές αποφάσεις. Καμία χώρα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα από μόνη της. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονίσει την εθνική απάντηση κάθε κράτους μέλους. Μπορούμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα και να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών ε, δεδομένων. Αλλά πρέπει να δράσουμε ως Ευρώπη, συλλογικά. Και θέλω να χαιρετήσω την εργασία της Λουξεμβούργιας και της Ολλανδικής Προεδρίας με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλη προτεραιότητα και για το Υπουργείο Ιστορικών και για το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι να προσεγγίσουμε την, ε, Τουρκία και να έχουμε καλύτερη αστυνομική συνεργασία και καλύτερη συνεργασία γενικότερα στο θέμα των εκδόσεων. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Μπορεί αυτό να είναι εντός, εκτός αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι εντός αρμοδιότητας των Ευρωπαίων Υπουργών υπευθύνων για τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια. Το σημαντικό είναι ότι γίνεται δουλειά από τις υπηρεσίες πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιτρομοκρατία. Έχουμε νέα εργαλεία που δεν είχαμε καν φανταστεί πριν από κάποια χρόνια. Και χαίρομαι γιατί αλλάζουν οι νοοτροπίες και σιγά σιγά πείθονται όλοι ότι η ανταλλαγή των πληροφοριών είναι απαραίτητη για την αντι, αντι, αντιτρομοκρατία, όπως ήδη η ανταλλαγή πληροφοριών είναι εξαιρετικά έντονη από τους τρομοκράτες μεταξύ τους ήδη. Βλέπετε ότι όλες αυτές οι εξελίξεις συγκλονίζουν τους πολίτες και υπάρχει ο πειρασμός να αναδεπλωθεί κανείς στα εσωτερικά του σύνορα και να επιστρέψει στην εθνική μόνο όραση των πραγμάτων. Και έτσι ε, είναι, αυξάνεται ο κίνδυνος για ρατσισμό, για ξενοφοβία και μπαίνει η εκάστοτε χώρα σε αυτό το φαύλο κύκλο. Κάτω το οποίο είναι πολύ δυστυχές και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε. Λίγες χώρες έχουν υποστεί τόσο βία η επίθεση από το διεθνή τύπο όσο το Βέλγιο. Θα ήθελα να σας επιθυμίσω την ε, επίθεση στο Ευρωπαϊκό στο Εβραϊκό Μουσείο στις Βρυξέλλες τον Μάιο. Ε, ο, ο, διεθνής τύπος ε, πραγματικά στυλίτευσε το Βέλγιο, όμως ο τρομοκράτης, εμείς τον βρήκαμε και δεν ήταν Βέλγος πολίτης, ούτε πέρασε μέσα από βελγικά σύνορα. Ενώ εμείς ως Βέλγιο ζητούσαμε εντονότερη συνεργασία μεταξύ των ε, εθνικών αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών για πάρα πολύ μεγάλο ε, χρονικό διάστημα. Στο Βερβιέ δύο τρομοκράτες βρήκαν το θάνατο. Μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι τεράστιες προσπάθειες κάναμε για να προχωρήσει η βελγική έρευνα και ανάκριση σε στενή συνεργασία ε, με τους Γάλλους μέσα από κοινέ ερευνητικές ομάδες. Οι Βέλγοι ερευνητές κατέβαλαν λοιπόν τεράστιες προσπάθειες και ε, σε συνεργασία με τους Γάλλους συναδέλφους κατάφεραν να εξαρθρώσουν αυτή ε, την ε, αυτή την ομάδα τρομοκρατών. Εξαρθρώθηκε και αποδυναμώθηκε και μόνο λίγα στοιχεία αυτής μπόρεσαν να κινηθούν τον, στις 22 Μαρτίου. Έχουμε Διερευνητική Επιτροπή στο Κοινοβούλιο που συγκροτήθηκε και θα εξετάσει τις ευθύνες σε όλα τα επίπεδα. Θα εξετάσει τις διαδικασίες και θα διατυπώσει συστάσεις ε, για βελτιώσεις όπου δει. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα είμαστε με τα κράτη-μέλη ε, τη πρώτη γραμμή για περισσότερη ολοκλήρωση, για περισσότερη ασφάλεια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων των ε, μελών του προσωπικού. Και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία και με τα λοιπά κράτη-μέλη σε επιχειρησιακό επίπεδο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους όσοι μας βοήθησαν στις δικές μας έρευνες από τις επιθέσεις στο Παρίσι και μετά αλλά και μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Σίγουρα πολλά μένει να γίνουν για να βελτιωθεί η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών. Όμως η ευρωπαϊκή ελληνική και ο κοινός αγώνας κατά της τρομοκρατίας δεν είναι κούφια λόγια, είναι καθημερινότητα. Καθημερινή πραγματικότητα για τους αστυνομικούς, τους εισαγγελείς, ε, τους δικαστικούς λειτουργούς μας. Συνάδελφοι, ε, ξέρετε ότι το Βέλγιο έχει συνηθίσει να του ασκείται κριτική και ξέρετε πολύ καλά ότι οι Βέλγοι αρέσκονται στο να επικρίνουν τους εαυτούς τους. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε επίσης το γεγονός ότι η βελγική κυβέρνηση πιστεύει ακρατάντως ότι το μέλλον βρίσκεται σε περισσότερη Ευρώπη και όχι σε λιγότερη. Δεν υπάρχει ε, δρόμος προς τα πίσω. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά όλο και πιο μπροστά ε, και με όλο και πιο ε, υψηλή ταχύτητα για να ε, καταπολεμήσουμε μία από τις πιο βάρβαρες πράξεις της εποχής μας που είναι η τρομοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πηγαίνουμε στην ανταλλαγή απόψεων ένα μέλος αναπολιτική ομάδα και μετά με σειρά χρονολογική προτεραιότητα. Δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ γιατί ο κύριος Ζαμπόν πρέπει να φύγει στις 4 και γι' αυτό άλλωστε ξεκινήσαμε τη συνεδρίαση στις 2.30. Παρακαλώ καλό να είστε επιθερχημένοι και να μην ε, ξεπερνάτε το χρόνο σας. Από το ΕΛΚ, ο κύριος Μπόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της ε, Κυβέρνησης ε, και Υπουργέ Δικαιοσύνης, καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω συλληπιτήριά μου, τα ελεπινή μου συλληπιτήρια από την πλευρά μα, και εμένα προσωπικά σε ό,τι αφορά αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις Βρυξέλλες. Νομίζω πως αυτή την περίοδο δεν θα πρέπει τώρα να προσπαθήσουμε να αποδίδουμε ευθύνε. Έχει φτάσει η ώρα να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το μέλλον και να δράσουμε από κοινού εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε την κοινή μα ασφάλεια. Και νομίζω πω για να το επιτύχουμε αυτό η λέξη κλειδί είναι η πρόληψη. Όπω έχουμε επαναλάβει πολλέ φορέ και στο παρελθόν Εκείνο που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι να υπάρχει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολή ε, του νόμου, των υπηρεσιών ε, πληροφοριών και των εμπλεκόμενων φορέων, όπω αναφέρθηκε από τον Υπουργό Κέντ. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να επιδεχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε την Ευρωπόλη, η οποία είναι σε θέση να κάνει πολλά περισσότερα εάν λαμβάνει γέρο τις κατάλληλες πληροφορίες. Δηλαδή το να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών είναι ένα πράγμα, αλλά από εκεί και μετά η επεξεργασία και η ανταλλαγή των επεξεργασμένων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο είναι κάτι ακόμα σημαντικότερο. Έχουμε την οδηγία για τα PNR, τα στοιχεία δηλαδή των επιβατών και αναμένουμε την ε, ε, θέση σε εφαρμογή και επίσης αναμένουμε την οδηγία για την ε, τρομοκρατία. Με αυτές τις νομοθετικές πράξεις θα έχουμε τα εργαλεία για να λαμβάνουμε πιο συγκεκριμένα ε, μέτρα ούτως ώστε να μπορέσουμε να ε, καταπολεμούμε αποτελεσματικά ήδη σε φάση την προετοιμασία της την τρομοκρατία. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε λοιπόν και ε, την ε, παρουσία των αλλοδαπών μαχητών και κατά συνέπεια θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτέ τι οδηγίε το ταχύτερο δυνατό. Επίση δεν θα πρέπει να ε, ξεχνούμε την πρόκληση που παρουσιάζει η ρίζο παστικοποίηση και εδώ θα πρέπει δηλαδή να ληφθούν μέτρα σε δημόσιο επίπεδο, τους, ώστε να αποφευθεί η ριζοσπαστικοποίηση και να διχθεί σε αυτά τα άτομα ότι υπάρχουν άλλε εναλλακτικέ. Θα πρέπει να ε, ε, δούμε πώ μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο του Darknet στην προώθηση αυτών των ομάδων ριζοσπαστικοποίηση. Αυτά και άλλα μέτρα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Αλλά να θέσω συγκεκριμένα ερωτήματα τώρα. Ε, τι νομίζετε πως χρειάζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από πρακτικής άποψης, ε, ποιες είναι οι δυναμίες τις οποίες εσείς εντοπίσατε σε ό,τι αφορά ε, στο επίπεδο της ε, ανταλλαγής πληροφοριών στην ε, πόλη των Βρυξελών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών. Επίσης, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την βελτίωση της ασφάλειας στο αεροδρόμιο του Ζάβεντεμ και στην ίδια την πόλη των Βρυξελών και πώς θα πρέπει μελλοντικά η συνεργασία να διαμορφωθεί ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες για την ασφάλεια που αναφέρθηκατε. Ευχαριστώ. για το S&D ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριοι Υπουργοί που είστε εδώ μαζί μας γιατί είστε μέλος ε, του Συμβουλίου Τζάι Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων και έχετε τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε. Θα ήθελα να σας υποβάλω ε, την εξής ερώτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Πιστεύω ότι είναι ο αδύναμος κρίκος. με ανησυχεί η τελευταία έκθεση σχετικά η οποία μας λέει ότι κάποιες χιλιάδες βρίσκονται μαχητές ε, στα αντίστοιχα μητρό και στις βάσεις δεδομένων, 5.000 κάτι, ενώ 1.600 γνωρίζουμε που βρίσκονται. Τους υπόλοιπους αγνοούμε που βρίσκονται. Λέτε λοιπόν ότι θέλετε να βελτιώσετε την ανταλλαγή πληροφοριών. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Εδώ και μήνες ε, μιλάτε γι' αυτό θα έχετε ένα οδικό χάρτη που θα αναθεωρείται ανατακτά χρονικά διαστήματα ε, με συγκεκριμένα στάδια που θα πρέπει να καλύπτονται για να ξέρουμε και ποιες χώρες προχωρούν και πόσο γρήγορα. Από εκεί και πέρα, ως προς τη Europol, τα κράτη-μέλη θα διαβιβάσουν τα στοιχεία στη Europol που χρειάζεται για να ε, διενεργεί στις αποστολές της. Το Βέλγιο θα το κάνει και τι θα κάνετε για να το κάνουν και οι υπόλοιπες ε, χώρες. Έχουμε την αντιτρομοκρατική υπηρεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ιδρύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες και όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να αποσπάσουν εκεί εμπειρογνώμονες. Το έχουν κάνει ή υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν το έχουν κάνει. Υπάρχουν τώρα κράτη-μέλη που δεν είναι συνδεδεμένα στο σύστημα σχένα της Ευρωπόλ και ό,τι έχει να κάνει με τους 3.000 περίπου ξένους μαρχητές που έχει η Europol στα αρχεία της έχει συμπεριλάβει την ταυτότητά του στη βάση δεδομένων Σέγγεν, του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. Δεν ψηφίσαμε την υποχρεωτική ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Αυτό το είχε προβλέψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά το Συμβούλιο ήταν όχι. Είπε όχι. Δεν θα έχουμε ένα PNR λοιπόν, ένα μητρό με τα δεδομένα των επιβατών, αλλά 28. Εσείς θέλετε να το εξαπλώσετε το PNR και να περιλάβετε εκεί και τις ε, σιδηροδρομικές και ε, θαλάσσιες μεταφορές. Πώς θα μπορέσετε να μεριμνήσετε για καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Όλοι ξέρουμε ότι αν δεν υπάρχει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, όσε βάσεις δεδομένων και να δημιουργήσουμε, δεν θα είναι και πολύ χρήσιμες. Ευχαριστώ. Για το ίσιο, ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εμείς από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Ε, θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν είναι πάντοτε αυτονόητο μετά από κάποιες τρομοκρατικές υποθέσεις οι συναρμόδιοι υπουργοί να προσέρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μας ενημερώνουν, αλλά το θεωρούμε πραγματικά πολύ θετικό και θα θέλαμε αυτό να ε, λαμβάνει η χώρα και γενικότερα με αυτόν τον τρόπο δηλαδή μπορεί να υπάρξει και ε, υψηλότερη πίεση προκειμένου να λαμβάνει χώρα εδώ ε, μια συζήτηση πάντοτε σε τέτοιε περιπτώσει, ώστε να μην περιορίζεται ο σχετικό διάλογο μόνο στο εθνικό επίπεδο. Άρα λοιπόν θεωρούμε πολύ θετικό το ότι ήρθατε σήμερα εδώ. Η η κυβέρνησή σας έχει πραγματικά εδώ ε, επιτύχει μια παράδοση εντός εισαγωγικών ε, ασφάλειας, ε, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να υποθεί για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά πραγματικά βλέπουμε ότι τώρα κάνετε σοβαρές προσπάθειες και βέβαια αυτές οι προσπάθειες εντοπίζονται και σε δύο επίπεδο, σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή σε διεθνές επίπεδο βλέπουμε ότι προσπαθείτε να ληφθούν μέτρα και σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη και μπορείτε να λειτουργήσετε ως υπόδειγμα εδώ, γιατί υπάρχουν εδώ και μήνες στρατιώτες οι οποίοι ε, προβαίνουν σε ε, ελέγχους και σε περιπολίες πράγμα ε, το οποίο ενδεχομένω θα μπορούσαν να εφαρμόσουν και άλλες χώρες. Επίσης στην παρουσίαση που κάνατε είπατε ότι δεν θέλετε να δημιουργήσετε ένα οποιοδήποτε σύστημα, αλλά θέλετε να έχετε πολύ, ένα σύστημα το οποίο θα είναι αποτελεσματικό, θα, θα έχει δηλαδή πολύ στοχευμένα μέτρα για να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όμως, σε ό,τι αφορά την ε, διαφοροποίηση ανάμεσα στο εθνικό και στο διεθνές επίπεδο. Μας είπατε ότι θέλετε ε, εδώ να κάνετε προσπάθειες και στα δύο επίπεδα. Μας είπατε ότι έχετε εστιάσει ειδικότερα στην πόλη των Βρυξελών, έχετε και συγκεκριμένα σχέδια εφαρμογή, αλλά από εκεί και μετά στο ευρωπαϊκό επίπεδο ε, μας είπατε ότι υπάρχουν κράτη μέλη τα οποία έχουν συνεργαστεί εντατικά μαζί σα και γνωρίζουμε ότι ο Υπουργό Διαμπών θέλει εδώ να προωθήσει περισσότερο αυτή τη συνεργασία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με αυτού του ε, υπουργού. Ναι, γνωρίζουμε ότι έλαβε χώρα ε, και η σε ό,τι αφορά το PNR, αλλά θα ήθελα να ακούσω τι πιο συγκεκριμένα θέλει ε, να συζητήσει ο Υπουργό την ερχόμενη εβδομάδα με του Υπουργού κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαμπόν, Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. διαπιστώνω άλλωστε ότι πρώτη φορά μετά από τρομοκρατική επίθεση καλούνται οι Υπουργοί να δώσουν εξηγήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και θαραλέο δεδομένου του τι βιώνει αυτή η χώρα σήμερα που ε, βρίσκεται στο στόχαστρο της διεθνούς ειδησιογραφίας η οποία συχνά θεωρεί ότι είναι η μόνη πηγή τρομοκρατών η χώρα του Βελγίου και λυπούμε πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να μιλήσω για τις ευθύνες των βελγικών αρχών. Έχετε, αρχών, έχετε υιοθετήσει πάρα πολλά μέτρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναγνωρίσει στην ε, ανακοίνωσή της. Πράγματι υπήρξαν κάποιες ανεπάρκειες στο βελγικό μηχανισμό. Ήμασταν σε κατάσταση συνεγερμού υπαριθμών 3 με την αστυνομία στους δρόμους, το στρατό κινητοποιημένο και ό,τι καταφέραμε το, ε, το κάναμε μετά. Το καταφέραμε μετά, όχι πριν. Δηλαδή μεταξύ Παρισιού και Βρυξελών θεωρώ ότι τα πράγματα δεν κινήθηκαν αρκετά γρήγορα και θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτή η περίοδος. Τώρα, για τις ιδιαίτερες ευθύνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι δύο επιμείνατε ιδιαίτερο στην ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία πράγματι ε, είναι ένα κέριο ζήτημα. Σήμερα μιλούμε για κοινό ορισμό των ξένων μαχητών, foreign fighters. Δεν έχουμε κοινό ορισμό για το τι είναι τρομοκράτης, ποιος είναι τρομοκράτης και ποια πράξη ακριβώς θεωρείται τρομοκρατική. Και θα έπρεπε για να έχουμε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ως προς τα PNR, δεν δέχτηκε το Συμβούλιο τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών. Συμφωνείτε εσεί οι δύο Υπουργοί με την απόφαση του Συμβουλίου, γιατί όταν θα είναι λειτουργικά και επιχειρησιακά τα PNR, οι τρομοκράτε και οι ξένοι μαχητέ θα πρέπει υποχρεωτικώς να γίνουν το αντικείμενο ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των μονάδων PNR των εθνικών υπηρεσιών των κρατών μελών, κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Εσεί είστε υπέρ αυτού του συστήματο. Αυτό καταρχάς, κατά δεύτερο λόγο. Ε, ε, επιχειρηματολογείται πολύ για υπέρ της συστηματικής συνεργασίας. Να σας ρωτήσω το εξής. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι σήμερα το 100% των ξένων μαχητών που απογράφονται στη βελγική επικράτεια έχουν ενταχθεί στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Είναι δεδομένο που έχει μπει στο σύστημα το 100% όσων έχετε εσείς εντοπίσει βρίσκονται μέσα στο SIS, το SIS. Και για την Ευρωπόλ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχει αντιτρομοκρατική πλέον υπηρεσία, μια μονάδα αντιτρομοκρατική η Ευρωπόλ. Έχετε κάποια στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συνεργασία σας με αυτή την υπηρεσία της Ευρωπόλ και αν ναι, υπό ποια μορφή γίνεται αυτή η συνεργασία. Ευχαριστώ. Η Λόρα Φεράρα για το EFTD παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τους υπουργού ε, που έχουν λάβει μέχρι τώρα το λόγο. Ευχαριστώ επίσης πολύ για όλα όσα κάνατε μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του αγώνα κατά της ε, τρομοκρατίας. Υπάρχουν βέβαια κάποια πράγματα τα οποία δεν επιστρέφουν και επ' αυτών θα ήθελα να έχω μία απάντηση. Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Τελικά τι δεν πήγε καλά. Μιλήσαμε για όλα αυτά που έγιναν εκ των υστέρων, την επομένη των τρομοκρατικών υποθέσεων. Όμως ξέρετε κάτι, εκείνο που δεν έχω καταλάβει καλά είναι τι έγινε εκ των προτέρων σε επίπεδο προληπτικό και τι δεν λειτουργήσε. Τι δεν πήγε καλά και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Αυτό που γνωρίζουμε και μας έχει ε, πλήξει όλους ήταν η έλλειψη προετοιμασίας. Έλλειψη προετοιμασίας ε, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και μάλιστα σε μια πόλη η οποία είναι η καρδιά της Ευρώπης. Παρά τις επιθέσεις στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Μαντρίτη, παρά ε, τη σύλληψη του Σαλά πριν από λίγες μόνο ημέρες, ε, θέλω να ρωτήσω, τι είναι εκείνο το οποίο δεν οδήγησε στο να ληφθούν κάποια μέτρα, παρότι υπήρχε κάποια ανησυχία. Υπήρχε ανησυχία και υπήρχε και η θέληση συνεργασίας ε, με τη δικαιοσύνη. Μήπως ξέφυγαν κάποιες πληροφορίες, ε, ε, δεν ήταν σωστές πληροφορίες, τι δεν πήγε καλά σε θέματα ασφάλειας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ τα συρρυκνώνω όλα αυτά σε μία πολύ απλή ερώτηση. Τι δεν πήγε καλά παρότι σας λέω είχαμε ήδη κάνει και κατά το παρελθόν παρεμπερίες εμπειρίες. Αυτό το ένα και κάτι άλλο πολύ πρακτικό. Εγώ εκείνη την ημέρα, εκείνη την περίφημη Τρίτη, πραγματικά ε, έφυγα τρέχοντας με το αυτοκίνητό μου προς την Ιταλία. Ξέρετε γιατί, δεν αισθανόμουν ασφαλής. Όπως και πολλοί άλλοι δεν αισθανόμουν ασφαλής να μείνουν ε, στο Βέλγιο. Και παρότι μας καλέσατε να μείνουμε στο σπίτι μας, να μην τα κινητούμε, εγώ έφυγα τρέχοντας. Και θέλω να σας πω ότι στη διαδρομή υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις στα σύνορα. Ε, λίγο μετά ε, τις επιθέσεις ε, υπήρχαν μεγάλες ουρές, αλλά ξέρετε κάτι, δεν υπήρχε καθόλου έλεγχος, ούτε έστω και συμβολικά, ένα αστυνομικό όχημα. Άρα δηλαδή όπως και εγώ που μπήκα στο αυτοκίνητό μου, και άρχισα να τρέχω να εγκαταλείψω όχι μόνο τις ε, Βρυξέλλες αλλά και το Βέλγιο γενικότερα, προφανώς το ίδιο θα μπορούσαν να έχουν κάνει και το Κάραν νομίζω και οι τρομοκράτε. Μα τελικά δεν καταλαβαίνω. Γιατί έστω και λίγες ώρες μετά την επίθεση δεν είχατε κανός είδους έλεγχο. Μιλήσατε για το Μητρό των Επιβατών, ε, για τη μεγαλύτερη συμβατότητα ανάμεσα στις ε, τράπεζες δεδομένων, κυρίως αυτές που έχουν στοιχεία των επιβατών. Υπάρχει τράπεζα δεδομένων του Σέγκεν, ε, υπάρχει τράπεζα δεδομένων για τα δακτυλικά αποτυπώματα, ε, τράπεζα δεδομένων της Europol, της Eurojust, κέντρο ευρωπαϊκό αντιτρομοκρατικό της Europol, ε, ένα άλλο κέντρο στο Συμβούλιο. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά εργαλεία και θεσμοί. Όμως κάθε φορά από ό,τι φαίνεται, εκείνο που δεν λειτουργεί καλά είναι η συνεργασία και η ανταλή, ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν υπάρχει η συμπατότητα που είναι απαραίτητη. Άρα, δηλαδή, καθαρά πρακτικά, τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Από το ΙΕΦΕΝ, e κυρία Μάγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια αίσθηση ντεζαβού. Γιατί μετά από κάθε τρομοκρατικό χτύπημα ε, ακούμε πάνω κάτω τα ίδια, δηλαδή βαρύγδουπες δηλώσεις, ε, τα κράτη-μέλη προτίθεται να λάβουν μια σειρά από μέτρα, αλλά τελικά ε, πάντοτε ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Και πραγματικά γίνονται κάπως αναξιόπιστα, όταν δηλαδή κανείς τελικά δεν θέλει να δει την αλήθεια κατάματα. Δηλαδή τα όσα συμβαίνουν αποτελούν τελικά συνέπεια της Ισλαμιστικής ιδεολογίας. Τα δικά μας σύνορα είναι ανοιχτά ε, και εγώ μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα ήμουν εδώ και ε, ταξίδεψα στις κάτω χώρες και δεν ε, πέρασα από κανένα είδου έλεγχο. Οπότε δεν βλέπω να υπάρχει κανένα είδου έλεγχο σε κάτι διαλευστό σύνορων. Οπότε αναρωτιέμαι τι έμαθε τελικά το Βέλγιο μετά από αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Και πώς το εξηγείτε εσείς ότι ο Σόλαμ Αμπτεσλάμ ε, ήταν σε θέση να ε, κρυφθεί για σειρά μηνών σε μια Ισλαμική κοινότητα στο ε, Μόλεμπεκ. Πώς μπορείτε λοιπόν να φροντίσετε για την ασφάλεια των πολιτών σας όταν δεν αναγνωρίσετε ότι το Ισλάμ αποτελεί τελικά την πηγή αυτού του φόβου. Να περάσω τώρα στα μέλη, ο πρόεδρος, ο κύριος Μισελ μπορεί να ξεκινήσει, παρακαλώ. Oui, euh... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργή, νομίζω ότι πρέπει να χαιρετήσω καταρχάς την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να είχαμε μπορέσει να προσκαλέσουμε επίσης και τους Γάλλους υπουργούς μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι. Υπάρχει θετική διάκριση λοιπόν υπέρ ημών με ύψιλον. Ίσως γιατί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες. Άγνωστο. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε ερωτήσεις και σε άλλους υπουργούς και όχι μόνο σε Βέλγους υπουργούς. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία σας εδώ είναι μια πολύ καλή ε, πρωτοβουλία. Υπάρχει Ερευνητική Επιτροπή που θα εργαστεί στο κοινοβούλιο στο Βέλγιο και μπορεί να διευκρινίσει τα πράγματα και ενδεχομένως η έκθεσή της να είναι πολύ πιο ενημερωτική για εμάς. Και δυστυχώς δεν μπορείτε να μας ενημερώσετε γιατί δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της η Επιτροπή αυτή και δεν έχει καταλήξει σε συγκεκριμένες συστάσεις. Ε, είναι υπό έρευνα λοιπόν το θέμα. Καταρχάς να πω ότι χαίρομαι γιατί ο φάκελος για το PNR, για τα μητρώα των ε, αεροπορικών επιβατών έχει τύχει έγκριση, έχει δοθεί συνέχεια σε αυτή την υπόθεση μετά από τόσους μήνες και εγώ είμαι απολύτως υπέρ ενός μόνου Ευρωπαϊκού Μητρώου Δεδομένων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών και όχι 28 διαφορετικών από τα 28 διαφορετικά κράτη-μέλη για να είναι ένα εργαλείο αποτελεσματικό. Και έτσι θα μπορέσουμε να επικεντρώσουμε τον ενδιαφέρον μας και τη δουλειά μας στα κριτήρια που θα καταστήσουν κάποιον ύποπτο ή μη. Σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον να συμφωνήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να ε, δουλέψουν πάνω σε αυτό το πεδίο, να έχουν κοινά κριτήρια, κοινέ παραμέτρους για να ξέρουν πώς θα εντοπίζουν ε, ε, τις ύποπτες ε, περιπτώσεις. Όσοι δεν θέλουν να προχωρήσουν να αφήσουν τους υπόλοιπους, δηλαδή να σημειώσουν την πρόοδο που, το που επιθυμούν. Μιλήσατε για τη βούλησή σας να καταπολεμήσετε τη ριζοσπαστικοποίηση, χωρίς βεβαίως να γίνονται γενικεύσεις και υπεραπλουστεύσεις. Ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι υπεραπλουστεύσεις, εξαιρετικά σοβαρό αυτό και άδικο και αντίκειται πλήρως στις ευρωπαϊκές αξίες και χαιρετίζω την κινητοποίησή την κινητοποίησή σας. Πράγματι το Βέλγιο κινήθηκε γρήγορα ενάντια της ριζοσπαστικοποίησης. Έγινε λόγος για ευρωπαϊκό Ισλάμ. Και κάθε θρησκεία που παρεκκλίνει από το κράτος δικαίου και που το θέτει σε κίνδυνο είναι για μένα επικίνδυνο. Όποια θρησκευτική ή πνευματική δύναμη υπάρχει που ε, θέλει να υπονομεύσει το κράτος δικαίου ή αντίκειται σε αυτό, αντιτάσσεται σε αυτό, για μένα είναι κάτι το επικίνδυνο ε, και θα πρέπει να ε, καταπολεμηθεί. Θα θέλαμε λοιπόν να μας διευκρινίσετε ε, όλες αυτές τις ερωτήσεις που έθεσα υπόψη σας. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, ε, να μπορέσει ο κύριος Γιαμπό να απαντήσει. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μην μακρηγορείτε. Η κυρία Σίπολ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, θερμά τους ε, υπουργούς ε, για την παρουσία τους σήμερα εδώ και θα ήθελα να πω παρά την ανασφάλεια που νιώσαμε μετά από τα τρομοκρατικά χτυπήματα εγώ αντέδρασα με διαφορετικό τρόπο δηλαδή και στις 22 του δεν επέστρεψα στην πατρίδα μου δηλαδή ήμουνα το απόγευμα στην πόλη των Βρυξελών και συνειδητά και αυτό βέβαια όπως σε πολλοί άλλοι ε, πολίτες ε, των Βρυξελών οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε κάπου αλλού για να κρυφτούν. Ε, και πέραν αυτού είχα βρεθεί και τα Χριστούγεννα, δηλαδή λίγο νωρίτερα στις Βρυξέλλες και να πω ότι πραγματικά σέβομαι το γεγονός ότι οι πολίτε ε, των ε, Βρυξελών παρά τα όσα πέρασαν ήταν διατεθειμένοι να ε, μην βρεθούν όμοιροι στην δική του την πόλη. Δηλαδή βγήκαν έξω στην πόλη και πραγματικά ήταν ε, μια αντίδραση την οποία σέβομαι και πραγματικά μια αντίδραση και δεν αναφέρομαι εδώ ε, σε εσά αλλά ε, την οποία δεν είδα από άλλους πολιτικούς γιατί βλέπουμε τελικά ότι πραγματικά όταν, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι προσπάθειες να υπάρχουν όλο ένα και πιο περιοριστικά μέτρα για να επιτύχουμε περισσότερη ασφάλεια, βλέπουμε ότι αυτό δεν πετυχαίνει πάντοτε θα πρέπει προφανώς να επανεξετάσουμε με κριτικό τρόπο τα ε, μέτρα ασφαλείας μας, από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ απόλυτη ασφάλεια. Οπότε ε, τέτοιου είδους τρομοκρατικά χτυπήματα όπως αυτά συνέβησαν στην ε, Γαλλία και εδώ στο Βέλγιο προφανώς υπάρχει η πιθανότητα να λάβουν χώρα. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι την κριτική που ασκήθηκε εδώ στο Βέλγιο, γιατί είμαι βέβαια ότι Αυτές, αυτή η κριτική που ασκήθηκε στο Βέλγιο ε, ισχύει και για άλλα ε, κράτη-μέλη τα οποία ε, δεν, στα οποία δεν ασκείται αυτή η κριτική μόνο και μόνο ακριβώς επειδή δεν έλαβε χώρα κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα. Κάτι το οποίο ε, επίσης με έχει εκνευρίσει στο πλαίσιο της όλου διαλόγου που γίνεται γύρω από την πολιτική ασφαλείας να πω ότι είναι το εξής. Όταν κανείς εξετάσει τα φαινόμενα αυτά της ρωσικοποίησης και τρομοκρατίας ε, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν μία σειρά από ε, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές ε, ε, αιτίες οι οποίες οδηγούν σε αυτό και ότι πάντοτε ε, τα ε, τρομοκρατικά χτυπήματα και η τρομοκρατία έχουν να κάνουν με την ε, μεταλλαγή των κοινωνικών παραμέτρων και γι' αυτό, γι αυτό τον, αυτή την πτυχή δεν άκουσα τίποτα σήμερα εδώ. Ο κύριο Ζαμπόν τώρα αναφέρθηκε σε 400 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διατεθούν για την ε, καταπολέμηση της νομοκρατίας εγώ θα ήθελα να μάθω ε, ποια είναι η κατανομή αυτών των ε, κονδυλίων, δηλαδή τι ακριβώς προβλέπετε για τη συλλογή των δεδομένων, τι προβλέπετε για τα μέτρα παρακολούθησης και ούτω καθεξής και τι κατευθύνεται στην μείωση της ριζοσυκοποίησης και στην πρόληψη, γιατί βέβαια και η πρόληψη αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε ολοένα και περισσότερους στρατολογούμενους. Και τέλος, κλείνοντας, να πω ότι υποστηρίζω πλήρως τα όσα είπε ο κύριος Μισελ δεν μας ωφελεί η συλλογή των δεδομένων όταν κάθε κράτος μέλος και κάθε εθνική υπηρεσία ε, προβαίνει ε, στην καταχώρηση αυτών των δεδομένων ε, και στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων με τελείως διαφορετικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση δεν μας ωφελεί η ανταλλαγή των δεδομένων γιατί ακριβώς δεν είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα μεταξύ τους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ακούσουμε τους όλους, γιατί η οι υπουργοί θα πρέπει να μα ε, να, να φύγουν. Οπότε οι τρεις επόμενοι ομιλητές, μόνο ένα λεπτό ο καθένας. Ο κύριος Μασούλα. Όχι, ε, πρόεδρε, έχω προσφέρει το δικό μου χρόνο αγόρευση στους συναδέλφους. Κύριος Μπέλη. Ευχαριστώ. Ένα έως δύο λεπτά, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ τους δύο υπουργούς για την παρουσία τους ε, σήμερα εδώ. Ε, τέθηκαν εδώ μία σειρά από ερωτήματα. Όπως για παράδειγμα το εάν θα μπορούσαμε να είχαμε αντιμετωπίσει εκπροβότερων και να αποφύγει αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα και τι ε, μπορεί να γίνει από εκεί και μετά. Ε, σίγουρα η απάντηση δεν είναι το να κλείσουμε τα σύνορα όπως προτάθηκε από μερικού εδώ. Δηλαδή κάτι τέτοιο εδώ είναι ανόητο και ανώφελο κιόλα. Οπότε θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η έμφαση να δοθεί στην πρόληψη και ταυτόχρονα και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Και όπω αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο, δηλαδή σε κάθε περίπτωση μπορώ να συμφωνήσω. Δεν ε, μπορούμε ποτέ να διασφαλίσουμε απόλυτη ασφάλεια. Όμω θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, ώστε να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιων χτυπημάτων. Και βέβαια εδώ ακριβώς εντάσσεται και η λογική της πολύ πιο αποτελεσματικής ανταλλαγής ε, των ε, πληροφοριών. Ε, το ιδανικό τι θα ήταν, ένα ευρωπαϊκού χαρακτήρα αν θέλετε FBI, αλλά βέβαια κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το επιτύχουμε, είναι μόνο ιδεατό. Οπότε σε αυτή τη φάση τι θα πρέπει να κάνουμε, να εστιάσουμε στα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία πραγματικά θέλουν να προχωρήσουμε περαιτέρω. Και αναφέρθηκε ήδη ε, ο κύριος Ζαμπών στο ζήτημα του συντονισμού ε, εκείνων των κρατών μελών τα οποία επιθυμούν να συνεργαστούν ε, εντατικότερο. Οπότε και σε σχέση με αυτό σας θέτω ένα ερώτημα. Θέλετε να λάβετε εσείς την πρωτοβουλία του ώστε από τη γαλλική κυβέρνηση και άλλα κράτη-μέλη για παράδειγμα να μαζευτούν 5-6 κράτη-μέλη τα οποία τελικά θα ξεκινήσουν αυτή την συνεργασία ούτως ώστε να υπάρξει τελικά ο πυρήνας εδώ μιας κοινή ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών. Ενδεχομένως δηλαδή να μην ξεκινήσει μια τέτοια υπηρεσία ευρωπαϊκού χαρακτήρα με 28 κράτη-μέλη, αλλά με 5-6 θα μπορούσε να γίνει η αρχή. Θα ήσασταν λοιπόν διατεθειμένο να αναλάβετε αυτή την πρωτοβουλία. Eh, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ε, δύο ε, υπουργού ε, από τη βελγική κυβέρνηση που ήρθαν σήμερα εδώ, ε, το είπαν και οι δυο ότι δηλαδή η καταπολέμηση της τρομοκρατίας έχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Οπότε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να να πούμε εδώ ότι αυτά τα μέτρα τα οποία είναι αποτελεσματικά και έχουν νόημα που έχει λάβει η βελγική κυβέρνηση να εφαρμοστούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει ε, να εστιάσουμε σε πολύ πρακτικά μέτρα. Ακούσαμε ούτω ή άλλω και από μια σειρά από ε, φιλελεύθερου εδώ συναδέλφου ε, ότι υποστηρίζουν τον, ε, τη δημιουργία ενό ευρωπαϊκού FBI και ενδεχομένω ακριβώ επειδή έχει δοθεί όθηση σε αυτή την πρωτοβουλία, ενδεχομένω θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε. Να υπάρξει δηλαδή μια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, αφού έχουμε και κοινά εξωτερικά σύνορα. Λέω, ε, ε, ακούσαμε επίση ότι θα υπάρξει μια περαιτέρω υποστήριξη, ενίσχυση τη Frontex. Μπορείτε να μα δώσετε περισσότερε πληροφορίε, τι ακριβώ ε, προβλέπετε. Σε κάθε περίπτωση όμω για να επιτευχθούν τέτοιου είδου μέτρα όπω ενίσχυση τη Frontex θα πρέπει να έχουμε και περισσότερη προσπάθεια από την πλευρά των κρατών μελών. Και η συνάδελφος που κάθεται ακριβώ πίσω μου να πω ότι ανέφερε ότι την ημέρα των τρομοκρατικών επιθέσεων έφυγε έντρομε από τις Βρυξέλλες ε, ε, ε, και πράγματι ένιωσα ότι υπήρξε αυτό το συνέστημα και σε άλλους εδώ, συναδέλφους και τελικά ε, ακούσαμε από κάποιους ε, στο Στρασβούργο ότι ενδεχομένως ε, θα πρέπει να συνεδριάζουμε εφ' εξής μόνο στο Στρασβούργο και να μην έχουμε ολομέλειες στο Κοινοβούλιο. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση αυτό που θα πρέπει να επιτύχουμε είναι από κοινού όλα τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν ούτως ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τις Βρυξέλλες και οι Βρυξέλλες να αποτελέσουν και πάλι μια πόλη στην οποία προσέρχονται όλοι ε, χαρά. So I go to Mr. John first. Ευχαριστούμε ε, όλους τους αδέλφους για αυτά τα λεπτομερά ερωτήματα. Ο κ. Ζαμπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ συναδελφοί για όλες τις ερωτήσεις που μου υποβάλλατε. Οι περισσότερες εξ αυτών ήταν πολύ κέρυες και Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μας αφορούν όλους και πρέπει να συνεργαστούμε για να τα αντιμετωπίσουμε. Πολλές ερωτήσεις ετέθησαν για την ανταλλαγή πληροφοριών, για το Μητρό των Επιβατών. Ε, θα τα απαντήσω όλα από κοινού και μετά θα πάω σε πιο μεμονωμένες ερωτήσεις. Όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων, ετέθη ένα ερώτημα, ε, κάποιος ρώτησε, ξέρετε ποια χώρα στέλνει πια δεδομένα. Στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνη, στο Τζάι, αποφασίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο κ. Κόβερ κάθε μήνα θα ε, μας παρουσιάσει την κατάσταση. Σήμερα έχουμε πληροφορίες μόνο όσον αφορά στη δική μας τη χώρα και μια γενικότερη εικόνα. Αποφασίσαμε όμως ότι το θέμα δεν είναι να ε, αποφεύγουμε να ονοματίσουμε. Το θέμα είναι να πείσουμε τις χώρες να δίνουν τα στοιχεία. Άρα δηλαδή τα στοιχεία θα διακινούνται στα Υπουργικά Συμβούλια και γενικότερα από την 1η Ιουνίου. Γιατί τώρα δεν έχουμε τις απαραίτητε πληροφορίες του ποια χώρα δίνει τις στοιχεία στη Europol. Σας λέω, από την 1η Ιουνίου όμως θα αλλάξουν τα πράγματα. Να σας πω επίσης ότι όταν μιλάμε για την παράδοση πληροφοριών στη Europol, το Βέλγιο είναι στην τρίτη θέση, αμέσως μετά τη Γαλλία και την Ολλανδία. Άρα δηλαδή νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όσον αφορά ένα άλλο σημαντικό θέμα για αυτούς που μετακινούνται, 611 εντοπίστηκαν οι ξένοι μαχητές, από εμά δηλαδή, αυτοί που πήγανε στη Συρία, κάποιοι πέθαναν, αλλά έχουν πληροφορίες και για άλλους που ετοιμάζονται να πάνε στη Συρία. Έχουμε όλες τις πληροφορίες για τους ε, ξένους μαχητές και αυτές τις δώσαμε. Έχουμε επίσης πληροφορίες για στρατολογητές και για συστήματα χρηματοδότησης. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε, όπως σας είπα, για ξένους μαχητές, για στρατολογητές και για την ε, χρηματοδότηση, για τα δίκτυα χρηματοδότηση. Εμείς τα έχουμε δώσει αυτά τα στοιχεία. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ε, όσον αφορά τη Europol, προφανώς είμαστε και υπέρ αυτής ε, και εμείς είμαστε και υπέρ της ε, πολιτικής ε, να ανταλλάσσουμε στοιχεία. Τώρα, ως προς μια κοινή ομάδα σύνδεσης με τη Europol. εξι κρατημέλη έχουν στείλει εμπειρογνώμονα και δύο που προτίθενται να το πράξουν. Άρα δηλαδή οκτώ κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Βελγίου. Ε, το Βέλγιο ήδη από τις είναι μία από τις έξι που έχει στείλει ένα εμπειρογνώμα σε αυτή την ε, κοινή ομάδα εμπειρογνωμόνων σύνδεσης. Κατόπιν τέτοιες ερωτήσεις για το PNR, αν είμαστε υπέρ ε, του, να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά το Μητρό Δεδομένων, ε, τους ξένους ε, μαχητές στο PNR. Κοιτάξτε, να πω το εξής, το ιδανικό θα ήταν να έχουμε ένα και σύστημα PNR. Αλλά πολλές φορές άλλο το ιδεατό και άλλο η πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ τάσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ του αυτό που έγινε, δηλαδή η Ολλανδία ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει πολλά κράτη-μέλη και να τα ε, πείσει να εφαρμόζουν το ίδιο σύστημα PNR. Αυτή την πρωτοβουλία την ανέλαβε η Ολλανδία και νομίζω ότι είναι μια καλή πρωτοβουλία γιατί ξέρετε κάτι θα έχουμε ένα ενιαίο σύστημα και σε μεταγενέστερη φάση θα μπορούμε περισσότεροι να πάμε σε αυτό το ένα και μοναδικό σύστημα. Καλή λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία της Ολλανδίας. Ως εκ τούτου, ναι, πράγματι, εγώ είμαι υπέρ της ανταλλαγής πληροφοριών. Υπάρχει ένας μαύρος κατάλογος ξένων μαχητών ε, που γνωρίζουμε και το εντοπίζουμε αυτό από τα διάφορα μητρώα δεδομένων και τα διαφορετικά συστήματα. Υπόθηκε να ε, περιλαμβάνουμε μητρώα και για τα τρένα. Όχι μόνο για τα αεροπλάνα. Να σας πω ότι στο δικό μας το πρόγραμμα προβλέπεται να υπάρχει ε, κατάλογος επιβατών όχι μόνο για τις ε, αεροπορικές μεταφορές αλλά και τις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές και για τα σκάφη και τα πλοία και για τα λεωφορεία γιατί υπάρχουν και πολλά λεωφορεία που μετακινούνται στην Ευρώπη. Κατ' ουσίαν το πρόβλημα είναι το ίδιο. Γιατί αν είμαστε εμεί ιδιαίτερα σκληροί με θέματα αεροπορικών μεταφορών, προφανώ και οι άνθρωποι αυτοί θα ε, βρουν κάποιε άλλε εναλλακτικέ λύσει ε, για να μετακινούνται. Νομίζω λοιπόν ότι απάντησα ε, σε αυτό το κομμάτι που αφορούσε την ανταλλαγή πληροφοριών και το PNR. Τώρα, να πάω σε άλλες ερωτήσεις. Νομίζω ε, τέτοι μία ερώτηση από εκπρόσωπο του ΕΛΚ ε, σχετικά με τις αδυναμίες στο δικό μας το, την αστυνομική διεύθυνση στις Βρυξέλλες. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι από αυτό. Αυτό είναι πολιτικής φύσης πρόβλημα στο Βέλγιο που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Κατά τη δική μου άποψη θα ήταν καλύτερο να έχουμε μία ζώνη, αλλά να σας πω κάτι, μερικοί δεν μιλάνε καν μεταξύ τους οι αστυνομικέ δυνάμεις. Έχουμε ένα συντονιστή για την πόλη των Βρυξελών που συντονίζει τις έξι ζώνες και μετά υπάρχει ανταλλαγή επιχειρήσεων, άρα το θέμα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Εγώ είμαι λοιπόν προφανώς και σίγουρος, αν είχαμε μία και μόνο αστυνομική ζώνη, ε, που θα περιλάμβανε και το Ζάβεντεμ και το Μάλμπεκ, τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Κατόπιν, με ρωτήσατε για την ασφάλεια στο αεροδρόμιο. Εκεί πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα ασφάλειας στο αεροδρόμιο και Πράγματι είναι πολλά, αλλά είχαμε να διαλέξουμε μεταξύ είτε αυτού είτε να μην ανοίξει καθόλου το αεροδρόμιο. Και τώρα, όταν θα ανοίξει το αεροδρόμιο στο σύνολό του, νομίζω ότι θα πρέπει να περιστεί και αυτή η περίμετρος ελέγχου. Γιατί ε, πράγματι δεν είναι αυτό δυνατό να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κύριε Λόνες, ε, με ρωτήσατε για το σχέδιο ε, του καναλιού. Είχε, αφορούσε στην αρχή το Μόλεμπεκ και τώρα αφορά ε, 7 ε, των Μεξελών και το Βιλβούρντε. υπάρχουν σχετικά κονδύλια που προβλέπονται για αυτήν την περιοχή. Αυτό το σχέδιο του καναλιού περιλαμβάνει δύο θέματα. Αφενό ένα ε, διοικητική φύσεως ε, σχέδιο, ένα άξονα διοικητικό, που σημαίνει ότι θα πρέπει ε, να υπάρχει καλύτερη καταγραφή από ό,τι κατά το παρελθόν. Δηλαδή θα καταγράφονται κάτοικοι του Μόλεμπεκ που ε, κατοικούν και όλες τις απαραίτητες άλλες λεπτομέρειες. Μετά, σε αστυνομικό επίπεδο, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εντοπίζουμε ε, αντιπαραθέσεις ε, στο Μόλεμε. Έχουμε 60 αστυνομικούς ε, για... Είχαμε 60 και τώρα θα τοποθετηθούν άλλοι 300 που θα δραστηριοποιούνται εκεί για να κάνουν σωστό έλεγχο θα ελέγχουν ας πούμε ε, τα πλαστά έγγραφα, διαβατήρια, αν υπάρχει αδιαπλοφορία, ε, τι γίνεται με τα ναρκωτικά. Αυτά θέλουμε όλα να ελέγξουμε σε αυτές τις περιοχές και γενικότερα το θέμα της μαύρης αγοράς. Ε, γιατί προφανώς και παίζει όλο και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. πόσον τώρα θα μπορούσε να υπάρχει μια μικρή μονάδα ε, για να ε, αναπτύσσει αυτά ταχύτατα και να αντιμετωπίζει ε, την τρομοκρατία. Μα την έχουμε αυτή. Είναι η ομάδα των 11 κρατών όπου βέβαια ευτυχώς δεν υπάρχουν και στα 28 κρατη τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι 11 όμως θεωρούν ότι ή είχαν ή θα έχουν, άρα δηλαδή γι' αυτό υπάρχει αυτή η ομάδα ταχύτατης δράσης και θέλουμε ε, να υπάρχει κάποια αρχή, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Ετέθη επίσης και ένα ερώτημα ε, σχετικά με την ε, Frontex, το προφίλ που θα πρέπει να εξετάζουμε. Κοιτάξτε, πρόκειται για συνοριακούς ελέγχους και εδώ πρέπει να υπάρχει στους συνοριακούς ελέγχους ένα ελάχιστο επίπεδο και νομίζω ότι ε, στο θέμα αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε. Κύριε Ντεπρέ, εσείς ρωτήσατε το εξής. Αν κάναμε τα πάντα μετά τις επιθέσεις που έπρεπε. Κοιτάξτε, στο Βερβιέ είχαμε λειτουργήσει ήδη πριν τις επιθέσεις. Μιλώ για τον Ιανουάριο του 2015. Την ε, δράση στο Βερβιέ την κάναμε τότε και μπορέσαμε να εντοπίσουμε την προετοιμασία όσους προ ετοιμάζονταν για αυτές τις πράξεις και εμείς θεωρούμασταν ήρωες, όχι εγώ προσωπικά βεβαίως, οι υπηρεσίες μας, οι άνθρωποι μας. Όλοι οι πρέσβεις στις Βρεξέλλες μου τηλεφώνησαν για να μου πούν πόσο καταπληκτική δουλειά έκαναν οι υπηρεσίες μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ηρωικές, παρόλο που οι πρέσβεις αυτό μου έλεγαν. Κάναν τη δουλειά τους, κάναμε τη δουλειά μας. Πιστεύω ότι οι υπηρεσίες μας είναι επαγγελματικές και η υπηρεσία πληροφοριών και η αστυνομική υπηρεσία. Είναι, έχουν υψηλό επαγγελματισμό, αλλά οι αντίπαλοι μας, οι τρομοκράτες, είναι επίσης επαγγελματίες. Είναι μηχανές πολεμικές έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά στη Συρία, γνωρίζουν πώς θα ανταλλάσσουν πληροφορίες ε, με διάφορους διάβλους επικοινωνίας σας ανέφερα ε, κάποιους στο διαδίκτυο είναι δουλειά, ε, είναι μια αρένα στην οποία από τη μία βρίσκονται επικελματίες και από την άλλη βρίσκονται επίσης επαγγελματίε να εγγυηθούμε 100% την ασφάλεια είναι κάτι που δεν γίνεται. Κανείς δεν μπορεί, καμία χώρα δεν μπορεί να πει σε όλους είστε 100% ασφαλείς. Μπορεί όμως να πει ότι θα κάνει τα πάντα για να προλάβει τις επιθέσεις και εμείς αυτό πράττουμε. Η αστυνομία μας, οι υπηρεσίε πληροφοριών, οι δικαστικές αρχές, οι εισαγγελικές αρχές δουλεύουν μέρα και νύχτα για να κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Δυστυχώς, ο μηδενικός κίνδυνος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος. Με ρωτήσατε σχετικά με το Ισλάμ. Κοιτάξτε, νομίζω το έχω πει εκατό φορές ότι το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή θα ήταν να καταστήσουμε το Ισλάμ εχθρό μας, πρότυπο εχθρού. Αυτό θα ήταν πραγματικά το χειρότερο. Στο Βέλγιο, ας πούμε, έχουμε περίπου 600-700.000 μουσουλμάνου και οι περισσότεροι εξ ε, είναι μουσουλμάνοι αλλά συμμεριζόνται τις ε, δικές μας τις αξίες. Αν λοιπόν όλους αυτούς τους ε, απορρίψουμε και τους πούμε είσαστε όλοι οι ίδιοι αυτό θα ήταν απόλυτα λάθος. Πρέπει να βρούμε ποιοι είναι οι τρομοκράτες και οφείλουμε τους μουσουλμάνους να τους καταστήσουμε συμμάχους μας αλλιώς θα υποπέσουμε σε μοιραίο λάθος. So Mr. Jeanbon will stay for a few minutes more and then he'll have to go. And I'm um, happy now to... Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να φύγετε σε λίγα λεπτά, οπότε να δώσω το λόγο στον Υπουργό κύριο Γιάννη, αλλά πρωτού ξεκινήσετε ε, να αναφερθώ σε αυτό που είπε και ο κύριος Ζαμπόν, ε, δηλαδή στις διακυβερνητικές ε, ε, συνεδριάσεις ε, και ε, ερωτήθηκα ότι αν ε, κάνουμε συνεντεύξεις αν θέλετε μόνο σε Βέλγους υπουργού. Ε, προφανώς ε, αντιλαμβάνεστε τον ειδικό χαρακτήρα της πρόσκλησης σας εδώ αλλά προφανώς θα προβούμε και σε συζητήσεις με άλλου υπουργού από και μετά το βασικό ερώτημα για μα είναι ε, το τι θα αποφασιστεί, τι θα εφαρμόσει στην πράξη δηλαδή το Συμβούλιο. Δηλαδή ακούμε να ε, συζητώνται όλε αυτέ οι προτάσεις ε, για ένα ευρωπαϊκό FBI και ούτω καθεξή. αλλά εκείνο που θα μπορούσε να βοηθήσει αυτή τη στιγμή το Βέλγιο είναι πολύ βασικές βάσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών. Για παράδειγμα, υπάρχουν και ήδη συμβάσεις εδώ, όπως αυτή του Προύμ, που θα μπορούσαν ακριβώς να βοηθήσουν, να συμβάλλουν στην ανταλλαγή των πληροφοριών. Οπότε, κύριε Χένσα, θα μπορούσατε να αναφέρετε τι θεωρείτε πως αυτή τη στιγμή λείπει. Γιατί βέβαια ο ρόλος μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το να εξετάζουμε ε, από πολύ κοντά τα όσα κάνει το Συμβούλιο και προφανώς και η Επιτροπή και να τους ε, θέτουμε ενώπιον των εθνικό γιατί προφανώ θέλουμε να σα βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε να πιάσετε του ε, τρομοκράτε. Ε, και σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη ε, ρησοπαστικοποίηση, ε, γνωρίζουμε ότι ε, συζητούνται πολλά και γίνονται πολλά, αλλά ε, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη είναι πολύ γενικά ε, και πολύ βασικά. Για παράδειγμα, ε, γίνεται η προσπάθεια κάποιων μέτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μέχρι στιγμή αυτά τα μέτρα δεν έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Οπότε θα ήθελα να σα ρωτήσω, ε, λαμβάνετε εσεί κάποια βοήθεια στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, γίνεται μια ανταλλαγή των πρακτικών, γιατί η πρόληψη αποτελεί πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, όλοι μιλάνε εδώ για την ριζοσπαστικοποίηση που λαμβάνει η χώρα στι δικέ μα χώρε. Και είναι κάτι το σημαντικό το οποίο βέβαια σχετίζεται και με την ε, ε, στη Συρία. Και εδώ βέβαια δεν αφορά αυτό το ερώτημα και αυτό το ζήτημα μόνο το Βέλγιο, αλλά και άλλε ευρωπαϊκέ ε, χώρε. Χένς, λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. επιτρέψτε μου να, να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα επιλεκτικά και συγκεκριμένα ξεκινώντας από το ζήτημα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και των αστυνομικών αρχών. Εγώ ε, προφανώς είμαι αρμόδιος ε, κυρίως για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ε, πληροφοριών και πολλά γίνονται μέσω τους ε, της Ευρωπόλ, αλλά υπάρχουν και άλλα επίπεδα. Για παράδειγμα υπάρχει το κλαμπ της Μπρον, το οποίο έχει, περιλαμβάνει και ένα ε, κομματικά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και χωρίς να, είμαι, να μην αποκαλύπτω όλα μυστικά εδώ, υπάρχουν πολύ βασικές διαστάσεις σε ό,τι αφορά τους ε, τρομοκράτες σε ε, ε, ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτές οι δύο πτυχές και τα σχετικά δεδομένα ανταλλάσσονται. Οπότε δεν θα πρέπει να θεωρούμε εδώ ότι δεν υπάρχει συνεργασία. Το ίδιο ισχύουν για παράδειγμα και το σύστημα SIS. Πολλές πληροφορίες ανταλλάσσονται και στο πλαίσιο αυτού του συστήματος και όπως Όμως είπε και ο Πρόεδρες, δυστυχώς συμβαίνει αναπεριόδους να υπάρξει μια κρίση για να θυμηθούμε ποιε είναι οι διεθνεί μα υποχρεώσει, όπω για παράδειγμα η διαβίβαση δεδομένων ε, στην Ευρωπόλ. Και όπω είπα, εμεί ανήκουμε στους, στα άριστα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την χορήγηση πληροφοριών στην Ευρωπόλ. Αλλά υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη που δεν το κάνουν. Και πραγματικά έχετε δίκιο όταν λέτε το Συμβούλιο ε, υπεύθυνο, αλλά και το Κοινοβούλιο. Είναι και περνάω εδώ σε ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό με το πρώτο, και αυτό είναι το εξή. Όταν αναφερόμαστε στην διατήρηση των δεδομένων, το, το PNR, τα στοιχεία των επιβατών, τον ορισμό της τομοκρατίας, εμείς δεν θεωρούμε ως Βέλγοι, δεν θα μιλήσω δηλαδή εξ ονόμαστου του Συμβουλίου, δεν νιώθουμε ότι λαμβάνουμε τη βοήθεια που χρειαζόμαστε. Και απαντώ ω Βέλγο γιατί ακριβώ τέθηκαν διάφορα ερωτήματα σαν να ήμασταν εμεί οι υπεύθυνοι για όλη την Ευρώπη. δεν συμβαίνει τίποτα σε επίπεδο για παράδειγμα ε, PNR. Έγιναν ε, προσπάθειες από την πλευρά του Συμβουλίου ε, και από την πλευρά τη Προεδρίας του Λουξεμβούργου, αλλά το Κοινοβούλιο δεν έκανε κάτι, ούτε η Επιτροπή έκανε κάτι. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για την πρωτοβουλία PNR. Δηλαδή, προφανώ ε, χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να ξεκινήσει και δεν αποτελεί αυτό μια αποτυχία για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά το Συμβούλιο. Το άκουσα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Επίση, θα ήθελα να πω κάτι ακόμα. Εγώ προέρχομαι από το ΕΛΚ. Έτσι, είμαι υπουργό τη βελική κυβέρνηση του ΕΛΚ, αλλά και αντιλαμβάνομαι ποια είναι η ιδιωτικότητα και προφανώ δεν είμαι υπέρ τη μαζική ε, παρακολούθηση. Υπάρχουν νόμοι στο Βέλγιο σε ό,τι αφορά την ιδιωτικότητα και τα όσα οι ε, δικαστέ θα πρέπει να σέβονται σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων για συγκεκριμένα πρόσωπα. Δηλαδή, για να υπάρξει μια συλλογή προσωπικών δεδομένων, πρέπει πάντοτε να παρεμβαίνει ένα δικαστή. Αλλά α μην είμαστε υπερβολικοί, για όνομα του Θεού, α μην είμαστε υπερβολικοί όταν έχουμε να κάνουμε με ζητήματα ασφαλεία. Είναι υπερβολικά περίπλοκα εδώ τα πράγματα και το είδαμε στην πράξη τι συμβαίνει. Οπότε, αναφερόμενος και πάλι σε αυτά τα δύο ζητήματα, στην διατήρηση των δεδομένων και ε, στα στοιχεία επιβατών ε, PNR, χρειάστηκε πολλής χρόνος και δεν φτάσαμε ακόμα στα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Ένα ακόμα ε, ζήτημα τώρα το οποίο θα ήθελα να θέσω. Και θα μιλήσω στα γαλλικά, γιατί με ρωτήσατε εσείς κυρία Φεράρα τι συνέβη και γιατί δεν δούλεψε το πράγμα. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ κύριε Φεράρα σε αυτό το ερώτημα. Είναι το αντικείμενο διερεύνησης της ε, ε, εξέτασης που κάνει το Βελγικό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω το εξής που ίσως ακουστεί ρητορία αλλά πρέπει να υποθεί. Είστε πολύ πιο νέα από μένα. Εγώ όμως περνούσα πάνω από τις μισές διακοπές μου στην Ιταλία εκείνη την εποχή, παρόλο που ήταν η περίοδος που δραστηριοποιούνται οι ερυθρές ταξιαρχίες. Μετά το αεροπλάνο που έπεσε στο Πεντάγωνο, μετά τα αεροπλάνα που έπεσαν στους δίδυμους πύργους, δεν είπε κανείς «δεν θα πάω στη Νέα Υόρκη» και την εγκατέλειψαν μαζικά. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο έχουμε αυτοκριτική και ίσως υπερβολική σε σύγκριση με άλλα κράτη και άλλα έθνη. Μην υπερβάλλετε. Ας μην υπερβάλλουμε γιατί δεν είναι λογικό. Εάν ένας άνθρωπος με ένα όπλο μπει σε οποιοδήποτε κτίριο, σε οποιαδήποτε πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη έχουμε πρόβλημα και δεν μπορούμε να κάνουμε πρόληψη 100%. 3.000 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στην Ευρώπη. Στη Νέα Υόρκη, με συγχωρείτε. Και δεν μπορούμε στην Ευρώπη να νομίζουμε ότι έχουμε το προνόμιο ότι θα γλιτώσουμε από όλο αυτόν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Πρέπει να είμαστε ε, σοβαροί, να σεβόμαστε τους εαυτούς μας. Και μάλιστα Έχετε δικαίωμα να ασκείτε κριτική βεβαίως. Εγώ ήμουν όμως στο κέντρο κρίσης και είδα από κοντά πώς γίνονται τα πράγματα. Εσείς μπορεί να μην είδατε κανένα στα σύνορα. Εμείς όμως στο κέντρο κρίσης αμέσως εποπτεύσαμε όλα τα σύνορα και τα γαλλοβέλγικα. Έχουμε πολύ περισσότερα σύνορα από ό,τι άλλες χώρες παρόλο που έχουμε μικρότερη γεωγραφική έκταση. Και κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Ο κύριος Μισελ μίλησε για το θέμα του Ισλάμ. Βεβαίως προσυπογράφω πλήρως ε, στα λεγόμενα του συναδέλφου Γιαμπών για το θέμα αυτό. Δεν θα πρέπει να δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Οφείλουμε όλοι στην Ευρώπη να συνειδητοποιήσουμε και ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ περισσότερους ε, ε, μουσουλμάνους παρά καθολικούς ή προτεστάντες στην Ευρώπη. Όχι μόνο γιατί είναι περισσότεροι μουσουλμάνοι, αλλά γιατί οι χριστιανοί είναι λιγότερο θρησκευόμενοι. Δεν πειράζει, δεν κακό αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα και οφείλουμε να τη γνωρίσουμε. Ε, έχουμε λοιπόν ε, μουσουλμάνους στη χώρα μας και έχουμε με με βασιλικό διάταγμα ε, ε βασιλικό διάταγμα τη σύσταση μιας εκτελεστικής ιεραρχίας που εκπροσωπεί τη μουσουλμανική κοινότητα στο Βέλγιο για να μπορούμε να διαβουλευόμαστε με εκπροσώπους αυτής της κοινότητας κάθε φορά που υπάρχει ε, λόγος. Εάν χρειαζόταν να έχουμε μια ομάδα, ένα εκτελεστικό σύστημα που να εκπροσωπεί τους χριστιανούς στο Βέλγιο, δεν θα ήταν τόσο απλό να συγκεντρωθούν εκπρόσωποι των χριστιανικών δογμάτων στην ίδια αίθουσα και να συμφωνήσουν συμφωνήσουν για την ιεραρχία μεταξύ τους και για το πώς και ποιοι θα είναι οι συνομιλητές του κράτους μας. Τα λέω όλα αυτά για να πω λοιπόν ότι ε, ρίζοσπαστικοποιούνται ορισμένοι από τους μουσουλμάνους. Η κοινότητα η τουρκική είναι υποδειγματική γιατί δεν παστικοποιείται. Όμως υπάρχει και πρόβλημα και με την τουρκική κοινότητα. Και προσπαθήσαμε να έχουμε ε, δημιουργία εκπροσώπων της τουρκικής ε, κοινότητας και δεν τα καταφέραμε και οι θύνοντες της τουρκικής κοινότητας προσέβαλαν την απόφαση που εξεδόθη με βασιλικό διάταγμα στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν λοιπόν, ε, υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία με την έννοια ότι ελέγχει τη διασπορά της, το, τους ε, Τούρκους του εξωτερικού και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν. Αυτά προς το παρόν κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Um, Κοιτάξτε ο Πρόεδρος, για τα θέματα του PNR θα έλεγα ότι είναι κάτι που ψηφίσαμε και για ένα μόνο νομοθετικό ζήτημα δεν θα έπρεπε να έχουμε τόσα πολλά σχόλια. Δεν ακούμε και πολλά για πολλές από τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Για αυτήν όμως την απόφαση έχουμε ακούσει εκατομμύρια πράγματα. Συμφωνώ μαζί σας. Το Βέλγιο ε, κάνει εισαγωγή των δεδομένων στα συστήματα της Ευρωπόλ. Όμως το Συμβούλιο δεν εφαρμόζει αυτά που χρειαζόμαστε. Όλοι ξέρουμε διαφάνεια τι έκανε το Κοινοβούλιο για το PNR. Και η κριτική που ασκήθηκε χαρακτηριζόταν από διαφάνεια, ήταν ανοιχτή και σαφής. Και αυτό θα ήθελα να πω. Νομίζω ότι κάνουμε παρατηρήσεις για την αντιριζοσπαστικοποίηση. Και όλα αυτά είναι χρήσιμα, αλλά έχει εξαντληθεί το θέμα σήμερα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε εδώ, ε, κύριε Υπουργοί. Ε, ήρθατε οικία τη Βουλήση και σας ευχαριστώ θερμότατα γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχετε συμβάλει στο να ε, προχωρήσει το ευρωπαϊκό έργο της ασφάλειας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά τους δύο υπουργούς της βελγικής κυβέρνησης καθώς και τα μέλη της Επιτροπής μας για αυτή την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Uh, if you're leaving. Συνάδελφοι, αν φύγετε από την Εύσο, παρακαλώ να φύγετε ησύχω. Θα πάμε ε, στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης και θα μας κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθύς αμέσως παρουσίαση για, την Ευρωπαϊ... για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ασφαλείας Καταπολέμησης Τρομοκρατίας και Δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη συνδέεται άρρηκτα με τη συζήτηση που είχαμε. Μιλώ για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε την περασμένη Τετάρτη για, την, για το πρόγραμμα, τη ημερήσια διάταξη για την ασφάλεια, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την διάνυση της απόστασης προς μια αποτελεσματική και πραγματική ένωση ασφάλειας. Κύριε Σορέκα, έχετε το λόγο. Στη συνέχεια θα γίνουν σχόλια και ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λουίτζι Σορέκα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που δίνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να παρουσιάσει αυτή τη σημαντική ανακοίνωση λίγες μέρες μετά την έγκριση αυτής της ε, πολιτικής. Είναι ένας χρόνος μετά τη θέση σε ισχύ της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ατζέντα για την ασφάλεια. Και τώρα έχουμε το πλαίσιο για το πώς θα δουλέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα για να πετύχει περισσότερη ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου και του σκέλους της τρομοκρατίας που μόλις τώρα συζητήσαμε. Το, οργανωμένο μένω έγκλημα και το κυβερνό έγκλημα και η τρομοκρατία είναι οι τρεις πυλώνες που πρέπει να καταπολεμήσουμε για περισσότερη ασφάλεια. Ένα χρόνο μετά την παρουσίαση της ατζέντα του πολιτικού αυτού προγράμματος είναι η κατάλληλη στιγμή σήμερα να κάνουμε έναν απολογισμό ότι έχει γίνει, ειδικότερα σε θέματα αντιτρομοκρατίας. Δεύτερον, να εντοπίσουμε κενά ε, στην εφαρμογή και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει εσάς ιδιαίτερα όπως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι η καλή στιγμή στιγμή να υπογραμμίσουμε ποιε δράσει φρονεί η Κομισιόν ότι χρειάζονται, δεν έχουν γίνει ακόμα για την καταπολέμηση τη ριζοσπαστικοποίηση. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τα υφιστάμενα εργαλεία για να έχουμε νέα δομή μεταξύ, και νέα συνεργασία μεταξύ των επιχειρησιακών υπηρεσιών που καταπολεμούν την τρομοκρατία. Και τέλος, η ανακοίνωση στέλνει ένα νέο και ισχυρό μήνυμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να προχωρήσουν προς τα εμπρός, πρέπει να προστατεύσουν την εσωτερική εθνική ασφάλεια. Η απειλή της τρομοκρατίας σε εθνικό επίπεδο ε, απειλεί την ασφάλεια της Ένωσης. Πρέπει να προστατεύσουμε τη συλλογική ασφάλεια της Ένωσης στο σύνολό της και αυτό πρέπει να γίνει ενάντια των πιο σοβαρών αδικημάτων, όπως είναι το αδίκημα της τρομοκρατίας. Η εσωτερική ασφάλεια ενός κράτους μέλους είναι εσωτερική ασφάλεια όλων των κρατών μελών. Και τα κράτη-μέλη είναι στην πρώτη γραμμή, είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια των, ε, της επικράτειάς τους. Αυτό προβλέπεται στη συνθήκη, αλλά δεν μπορεί κανένα κράτος μέλος να δράσει μόνο του και γι' αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να διαμορφωθούν τα εργαλεία, να οικοδομηθεί η υποδομή να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο οι εθνικές αρχές θα δίνανται να δουλέψουν και να αντιμετωπίσουν από κοινού προκλήσεις όπως η τρομοκρατία. Αυτό άλλωστε εννοούσε ο πρόεδρος Γιούνκερ όταν πήρε το λόγο στην Ολομέλεια και μίλησε για μια αποτελεσματική και λειτουργική πραγματική ένωση ασφαλείας όπου οι ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών θα τη χάνουν της επαρκούς προστασίας. Επιταχύνουμε την ε, εφαρμογή της ε, ατζέντα αυτής της πολιτικής και θα πρέπει η Επιτροπή σας να εξετάσει λοιπόν την οδηγία για την τρομοκρατία, την οδηγία για την, ε, ε, την απόκτηση και χρήση των πυροβόλων όπλων, την οδηγία για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης ε, Ποινικών Μητρών, έκρης και διάφορα άλλα θέματα. Έχει σημειωθεί πρόοδος και θα πρέπει να εστιάσω τον, το ενδιαφέρον μου σε τέσσερα ζητήματα. Αυτά τα τέσσερα ζητήματα αναδεικνύουν το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, η εφαρμογή, η υλοποίηση, το αναφέρατε και εσείς στις παρατηρήσεις σας. Πέρσι, ε, από πέρσι έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές πρωτοβουλίες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Νέα εργαλεία που προσθέτουν στο σύστημα, φέρνουν τη θεμενή αξία, αλλά δεν εφαρμόζονται πλήρως πάντοτε. Έχει έρθει η ώρα να δράσουμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει ασκή τις αρμοδιότητες που τις προβλέπονται από τη συνθήκη για να διασφαλίσει την εύρυθμη εφαρμογή και υλοποίηση από τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, ε, ανταλλαγή πληροφοριών. Αναφέρθηκε και νωρίτερα. Τρομοκράτε που είναι γνωστοί στη μία χώρα δεν θα πρέπει να διαφεύγουν του εντοπισμού στην άλλη χώρα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει διάφορες δράσεις για να βελτιώσει την ανταλλαγή των πληροφοριών. Όμως, όπως συζητήσαμε και προλίγου, χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες σε θέματα διασύνδεσης, διαλειτουργικότητας των διαφόρων συστημάτων που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Τρίτον, κοινή αξιολόγηση απειλών για να συνεργαστούμε καλύτερα και να καταπολεμήσουμε καλύτερα την τρομοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να έχουμε κοινή αντίληψη των απειλών και των κινδύνων. Το κατακαιρματισμένο τοπίο δεν επιτρέπει τη συντονισμένη απάντηση. Καλή δουλειά κάνει η Ευρωπόλ, καλή δουλειά κάνουν τα κέντρα, τα ίνσεν, τα εθνικά κέντρα ε, υπηρεσιών πληροφόρησης και συλλέγουν τις πληροφορίες και κάνουν αναλύσεις. Πρέπει να συγκεράσουμε όλη αυτή την εμπειρογνωμοσύνη του κάθε κράτους μέλους κοινή αξιολόγηση απειλών, ρίζοσπαστικοποίησης. Ε, αυτή είναι μια δραστηριότητα που κάνει το ECTC της Ευρωπόλ. Τέταρτον, πυροβόλα όπλα. Πρέπει να περικόψουμε την πρόσβαση των τρομοκρατών στους εκρηκτικούς μηχανισμούς, τους πυροδι πυροδοτικούς μηχανισμούς στα πυροβόλα όπλα. Ε, αυτό το μήνα ξεκίνησαν να ισχύουν νέοι κανόνες και αυτό μας ικανοποιεί. Έχουμε υποβάλει μια νέα πρόταση για τον έλεγχο και την κτήση των πυροβόλων όπλων, την αγορά όλων αυτών για το πώς ελέγχουμε καλύτερα την αγορά τους. Δεν αρκούν όμως αυτά. Υπάρχουν κενά στην εφαρμογή ε, της νομοθεσίας για τον εντοπισμό των πρόδρομων ουσιών, αν θέλετε, υλικών που μπορούν να, εύκολα να γίνουν εκρηκτικά υλικά και συστατικά στοιχεία του εκρηκτικού μηχανισμού. Ότι είναι δηλαδή οι πρόδρομες ουσίες ε, σε σχέση με τα ναρκωτικά είναι υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια να αγοραστούν και να τα αποκτήσει κανείς ε, και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσει για να φτιάξει εκρηκτικό και πυροδοτικό μηχανισμό. Ε, σε κάθε περίπτωση είναι κοινή ευθύνη και πρέπει όλοι να κάνουν αυτό που τους αναλογεί για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών και για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όλες αυτές οι απειλές. Και θα πρέπει οι διοκτικές αρχές, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών να συνεργαστούν, να ενώσουν τους πόρους τους ε, για να υπάρξει αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο Πρόεδρος, ευχαριστώ Λουίτσι. Αυτά δημοσιεύθηκαν την περασμένη Τετάρτη, συνάδελφοι. Είναι εξαιρετικά σημαντικά δεν ξέρω όμως αν είχατε την ευκαιρία να τα εξετάσετε ε, λεπτομερώς. Αν όχι, ο κύριος Λουίτζη σε κόρα μόλις σας έκανε μια πολύ χρήσιμη σύνοψη και τονίζεται πόσο σημαντική είναι αυτή η ανακοίνωση. Επομένως, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη που παρίστανται Θέλει κάποιος το λόγο. Ο κύριος Χάρλε Χαρφό για τα πυροβόλα όπλα φαντάζομαι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία αυτή η ανακοίνωση. Απλώς ε, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στο σύριο δράση για τα πυροβόλα όπλα και τα εκρηκτικά, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ε, προτινόμενη νέα οδηγία για τα πυροβόλα όπλα που έχει τεθεί προ και εδώ σε αυτή την Επιτροπή και γενικότερα στην Ευρώπη έχει καταστεί σαφές ότι πολλά από τα όσα προτείνονται στις, από την πλευρά της Επιτροπής δεν έχουν να κάνουν με την τρομοκρατία γενικότερα με εγκλήματα που σχετίζονται με όπλα, αλλά πρόκειται για μια ιδεολογική, ε, αν θέλετε, καμπάνια εκστρατεία κατά της ε, νόμιμης κατοχής ε, όπλων. και μάλιστα στρέφεται κατά των, νομίμων νόμιμων όπλων παρότι όσα έχουν χρησιμοποιηθεί από τρομοκράτε ήταν πάντοτε παράνομα και βλέπουμε ότι να υπάρχει μια ε, πρόθεση να τιμωρηθούν οι ε, κάτοχοι νομίνουμων όπλων μόνο και μόνο ούτως ώστε να ε, τους τιμωρήσουν για τις δικές τους αποτυχίες, δηλαδή την μη επαρκή καταπολέμηση τη τρομοκρατίας. Επίσης, με πολύ κοινικό τρόπο η Επιτροπή ε, έχει προσπαθήσει να αξιοποιήσει τον πανικό μετά από τα τρομοκρατικά χτυπήματα ε, του Παρισίου ε, προκειμένου να προωθήσει τη δική της πρόταση, η οποία βέβαια δεν πληρεί τα ίδια τα προαπαιτούμενα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον εαυτό του σε ό,τι αφορά την καλή νομοπαραγωγή. Οπότε, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Ε, ευχαριστώ. Πράγματι δεν είναι ε, εύκολο να εξετάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σε λεπτομέρειες, οπότε θα ήθελα να τονίσω εδώ το ότι ε, το να προσπαθούμε να πιέζουμε τα πράγματα και να είμαστε όσο το δυνατό ταχύτεροι ε, δεν είναι πάντα το καλύτερο σύμβουλο αν θέλουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Ε, πριν από λίγο ο Υπουργό Δικαιοσύνη μα είπε ότι όταν κάνουμε λόγο για νέα μέτρα ασφαλεία δεν θα πρέπει να δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση σε ζητήματα ε, ε, ιδιωτικότητα και προστασία των δεδομένων. Όμω νομίζω πω μπορούμε να πούμε και το αντίστροφο, δηλαδή ότι ε, όταν προσπαθούμε να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και αντίστοιχα μέτρα να πηγαίνουμε ε, πολύ μακριά. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί μετά από τα τρομοκρατικά χτυπήματα έχουν ε, τεθεί επιτάπητος μία σειρά από διαφορετικές ε, προτάσεις. Οπότε το δικό μου ερώτημα είναι, εάν υποθέσουμε ότι θα εφαρμοστούν σε κάποια ε, στιγμή όλα αυτά τα μέτρα και λάβει χώρα ένα ακόμα τρομοκρατικό χτύπημα. Τι θα σκαρφιστούμε αν θέλετε ε, παραπάνω τόσο ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερη παρακολούθηση, ακόμα περισσότερο έλεγχο των πολιτών μας. Και με απασχολεί λίγο το γεγονός ότι κάνουμε λόγο για μία σειρά από νέα μέτρα, αλλά ταυτόχρονα ακούμε ότι τα όσα ήδη εφαρμόζονται, τα όσα ήδη υπάρχουν, δεν εφαρμόζονται πλήρως, δεν εφαρμόζονται σωστά. Οπότε ενδεχομένω κάποια από τα νέα μέτρα να μην είναι απαραίτητα ή να μην ήταν απαραίτητα εάν εφαρμόζαμε με σωστό τρόπο τα όσα ήδη έχουμε στη διάθεσή μας. Οπότε φοβούμε ότι υπερβάλλουμε λίγο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό FBI όπως αναφέρεται, εγώ έχω να θέσω ένα απλό ερώτημα. Από όσα εγώ κατάλαβα, το FBI αποτελεί μια πρωτίστως πολιτική οργάνωση ε, η φορέα. Αλλά τώρα λέμε ότι ουσιαστικά θα είναι μια μυστική υπηρεσία η οποία θα ε, ε, διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατομελών. Οπότε τελικά τι θα είναι. Θα είναι ένας πραγματικά πολιτικός φορέας για τη συνεργασία μεταξύ των κρατομελών... ή ένας αστυνομικού χαρακτήρα φορέας. Αλλά ό,τι και αν αποφασίσουμε, ε, το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα έχουμε ε, ένα ε, ευρωπαϊκό FBI που θα αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση χωρίς να έχουμε κοινούς κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το τι επιτρέπεται να κάνει μια αστυνομική αρχή, τι δεν επιτρέπεται να κάνει, ποια είναι τα δικαιώματα των υπόπτων ή κατηγορουμένων. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο, πώς μπορούμε να μιλάμε για μια ένα κοινό αστυνομικό φορέα. Αυτό δηλαδή μου φαίνεται πως είναι ένα δεύτερο βήμα, το οποίο όμως θα έπρεπε να ακολουθήσει μετά από το πρώτο που είναι ακριβώς ένα κοινό πλαίσιο. Τώρα σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, νομίζω πως δεν έχει νόημα να αποστέλουμε κάποια κράτη-μέλη από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Έτσι απλά. Λέγοντα δηλαδή το ένα κράτο μέλο στο άλλο, πάρτε τα κάτω ό,τι θέλετε με αυτά τα δεδομένα. Χρειάζεται κανεί να ερμηνεύσει κατά κάποιο τρόπο αυτά τα δεδομένα. Και αυτό σημαίνει τι συνάντηση μεταξύ διαφορετικών εμπειρογνωμών των διαφόρων κρατών μελών, ούτως ώστε να υπάρχει σωστή ερμηνεία αυτών των δεδομένων. Και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό από την απλή ανταλλαγή των πληροφοριών, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες σκέψεις και να έχει, γιατί σε διαφορετική περίπτωση απλώς θα έχουμε ε, ε, συνέπειες για τους αυτούς πολίτες μας. Ε, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ακριβώς για οποιουσδήποτε παρακολουθούν μέσω web streaming αυτή τη συνεδρίαση. Να πούμε ότι σε αυτήν εδώ την ανακοίνωση της Επιτροπής δεν αναφέρεται κανένα ευρωπαϊκό FBI με κανένα τρόπο. Οπότε, εντάξει, μας λέτε ότι σας εκνευρίζει απλά αυτή η πρόταση, αυτό το ζήτημα του Ευρωπαϊκού FBI, αλλά εγώ απλώς να αναφέρω ότι αναφέρθηκε ούτως ή και στην προηγούμενη συνεδρίαση και υπάρχουν πολύ σημαντικά ερωτήματα γύρω από αυτά. Απλώς διευκρινίζω ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής δεν αναφέρεται κάτι σε σχέση με ένα ευρωπαϊκό FBI. Το επενθυμίζω απλώς αυτά. Κατρίνα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για αυτή την παρουσίαση. Πραγματικά έγινε λόγο για αυτό το ε, εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα τη ε, τρομοκρατία και σε διεθνέ επίπεδο και θα πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα και σε νομοθετικό επίπεδο, στο επίπεδο τη επιχειρησιακή δράση και ούτω καθεξή. Και βέβαια εδώ συγκαταλέγεται η ανταλλαγή των πληροφοριών και ο συντονισμό μεταξύ των αστυνομικών αρχών των και των δικαστικών αρχών, αλλά θεωρώ πως εξίσου σημαντικό είναι να δοθεί έμφαση στην διάσταση της ε, πρόληψης, ε, δηλαδή σε ό,τι αφορά την, ε, το profiling, την ανάπτυξη προφίλ δηλαδή και από εκεί και μετά βέβαια να, να εξεταστεί και το ζήτημα ειδικότερα της περιθωριοποίησης. Δηλαδή όταν κάποιος περιθωριοποιείται τότε είναι πολύ πιθανότερο να χρησιμοποιήσει και βία μέσα, ειδικότερα όταν μιλάμε για εφήβους και νέους ενήλικες. Επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε ειδικότερα με το ζήτημα ε, της ριζοσπαστικοποίησης στις ε, φυλακές ασοφρονιστικά καταστήματα. Αλλά από εκεί και μετά υπάρχει και ένα ακόμα θεματικό πεδίο στο οποίο δεν έχουμε αναφερθεί ιδιαίτερα, ε, το οποίο είναι η πρόληψη στο επίπεδο του διαδικτύου, γιατί υπάρχουν ακριβώς αυτά τα νέα μέσα επικοινωνίας και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η στρατολόγηση ατόμων γίνεται και μέσω του διαδικτύου. Και για παράδειγμα ότι μέσω του διαδικτύου μπορεί κανείς να φορτώσει στο σύστημά του τις οδηγίε χρήση για το πώ μπορεί να παρασκευάσει ένα εκρητικό μηχανισμό. Οπότε θα πρέπει να δούμε εδώ πώ μπορούμε να συνεργαστούμε και ε, με τους ε, με τις επιχειρήσεις σε αυτό το τομέα και με την Ευρωπόλη, ώστε να επιτύχουμε ε, την απομάκρυνση τέτοιου είδους περιεχομένου από το διαδίκτυο. Κάτι τέτοιο δηλαδή θα πρέπει να είναι δυνατό να γίνει. γιατί αποτελεί και αυτό ένα αποτελεσματικό τρόπο για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Επίσης θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση η οποία είναι ιδιαίτερα περιπλοκή. Δηλαδή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι προφανώς όλοι χαίρουν του δικαιώματος της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε σχετικές πληροφορίες. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις του κλάδου, ούτως ώστε να επιτύχουμε κάτι και σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να διατηρήσουμε προφανώ την ελευθερία στην πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά ταυτόχρονα να απομακρύνουμε τέτοιο περιεχόμενο έτσι ώστε να ε, προλάβουμε την τρομοκρατία που προωθείται και μέσα του διαδικτύου. Πρόεδρος. Ναι. Σε ό,τι αφορά αυτό το ε, σοβαρό ζήτημα που αναφέρθηκε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή στην πράξη. Αν ε, δούμε την ανακοίνωση θα δούμε ότι από το δεύτερο ε, τρίμηνο του 2016 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2017 έχουμε 17 διαφορετικές πολιτικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες και αθεωρήσεις πολιτικής. Οπότε το ερώτημα που εγώ θέτω είναι όταν λέτε όταν ε, κάνετε λόγο για εφαρμογή, αναφέρεστε σε δύο πράγματα. Δηλαδή, εφαρμογή σα νομοθεσία. και υπάρχει ακριβώς εδώ ε, η υφιστάμενη νομοθεσία για την οποία χρειαζόμαστε περαιτέρω ε, μέτρα και συμπληρωματικά ακριβώς αυτή η τα επιπρόσθετα μέτρα στο πλαίσιο της ισχύωσης νομοθεσίας. Το δεύτερο κομμάτι, η δεύτερη δηλαδή διάσταση της εφαρμογής, είναι η εφαρμογή των όσων ακόμα δεν λαμβάνουν χώρα ε, στο, ε, μέχρι στιγμής για παράδειγμα ανταλλαγή πληροφοριών, διατήρηση στο δεδομένων και ούτω καθεξής. Οπότε ε, ε ρωτάω αυτή η δεύτερη διάσταση σκοπεύετε να, την, να της δώσετε περισσότερη έμφαση μέσα σε αυτήν την ανακοίνωση ούτως ώστε να είναι σαφέ αυτό και για τους πολίτες και επαναλαμβάνω έχουμε δύο είδη ε, ε, εφαρμογή, επιβολή Δηλαδή, από τη μία έχουμε υφιστάμενη ισχύουσα νομοθεσία και από την άλλη ε, συμπληρωματικά μέτρα. Προφανώ χρειαζόμαστε ε, περισσότερη δηλαδή νομοθεσία σε ό,τι αφορά ε, την ατζέντα για την ασφάλεια, το γενικότερο θεματολόγιο, αλλά από εκεί και μετά υπάρχει και νομοθεσία και θα πρέπει να γίνει και μια αξιολόγηση της ε, σε διαφορετική περίπτωση. Αυτή η ανακοίνωση το μόνο που θα προβλέπει είναι τελικά περισσότερο φόρτο εργασίας για μας. Θα πρέπει λοιπόν να το κοιτάξετε και αυτό το ζήτημα ούτως ώστε να έχει προσθέμενη αξία αυτή η ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τους βουλευτές ε, κατανοώ βέβαια ότι δεν είχατε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το κείμενο, το οποίο, όπως σας είπα, έχει τρεις διαστάσεις και ίσως είναι και πιο φιλόδοξο από ό,τι θα ήθελαν μερικοί. Το μήνυμα που θέλω να περάσω ε, στην εισαγωγή μου αυτή είναι ε, και αυτό πολιτικά φιλόδοξο και ελπίζω ότι αυτό θα το λάβουν υπόψη τους οι, πολιτικές, ε, οι πολιτικά αρμόδιοι στην Επιτροπή. Θα ήθελα τώρα να προσπαθήσω να σας εξηγήσω περισσότερο την ουσία της ερώτησής σας και ξεκινώ με την ερώτηση της κυρίας Σίπελ σχετικά με το κατά πόσον από τη στιγμή που όλα τα μέτρα που έχουμε λάβει υπόψη μας εφαρμοστούν στην πράξη, κατά πόσον θα μπορούμε με τον τρόπο αυτό να αποφύγουμε άλλη μία τρομοκρατική επίθεση. Ε, η ασφάλεια, πρέπει να πω, ποτέ δεν μπορεί να είναι 100% και κατά δεύτερον δεν υπάρχει πλήρης εφαρμογή των μέτρων. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε το κατά πόσον τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει είναι αποτελεσματικά ή όχι. Γιατί όπως αναφέρει και η ανακοίνωση δεν υπάρχει πλήρης εφαρμογή των προτινόμενων μέτρων. Ούτε και αυτά που ελήφθησαν ε, εφαρμόζονται κατά 100% όπως είχαν προβλεφθεί. Ο πρόεδρος κύριος Μωράες ε, ρώτησε πότε η Κομισιόν θα καταθέσει νέες προτάσεις και κατά πόσον η Κομισιόν θα κάνει τη δική της αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή. Η απάντηση είναι προφανώς ε, και θα γίνει δική μας αξιολόγηση. Υπάρχει ένας ολόκληρος ε, κατάλογος μέτρων που αναφέρονται στο παράρτημα και όλα αυτά έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών. Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα δράσης που δημοσιεύτηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, πολλά εξ αυτών των μέτρων ήδη προβλέπονται, βρισκόνται σε φάση προετοιμασίας και ε, μία μελέτη αξιολόγησης ε, θα υποβληθεί μαζί με προτάσεις που θα αφορούν στην αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας θα περιλαμβάνουν μια αναθεώρηση οδηγίας περί ε, παγώματος ε, κεφαλαίων και κατάσχεσης ε, περιουσιακών στοιχείων. Πράγματα θα λοιπόν μια τέτοια σχετική πρόταση. Τώρα όσον αφορά τις, τη δραστηριοποίηση, η δική μου επιτροπή έχει τοποθετηθεί επ' αυτού με απόλυτη σαφήνεια. Και όπως σας είπα στην εισαγωγή μου έχουμε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες που έχουμε σε περιπτώσεις παραβίασης, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η μη εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών θα αντιμετωπιστεί. Δεν χρειάζεται να επανέλθω στο Ευρωπαϊκό FBI. Ε, παραλαμβάνω αυτό δεν αναφέρεται στην ανακοίνωσή μας και έχοντας κατά νου ε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο μετακινούμεθα, η Κομισιόν δεν έχει καμία πρόθεση να αλλάξει οτιδήποτε. Όσον αφορά την ενημέρωση, κυρία Σίπελ, πολύ σωστά επισημάνατε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ε, τεχνογνωσία των κρατών μελών. Και αυτό προτιθέμεθα να το κάνουμε, συστήνοντας μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη, αλλά και από άλλους εμπειρογνώμονε, από τον ιδιωτικό τομέα, ακαδημαϊκούς και αυτά όλα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της ε, διαλειτουργικότητας. Όλες αυτές οι ομάδες θα έχουν εμπειρογνώμονες, όπως σας είπα, από τα κρατη θα καταθέτουν προτάσεις στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο, πριν ε, λαμβάνονται δράσεις ε, για ε, δραστηριοποίηση. Ο κ. Κινίτσιο αναφέρθηκε στην πρόληψη. Βλέπω ότι εσείς είχατε τελικά χρόνο να διαβάσετε την ανακοίνωση και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Διαπιστώσατε ότι υπάρχει μια ειδική αναφορά στη ρίζοσπαστικοποίηση στις φυλακές. Υπάρχει ένα κεφάλαιο ολόκληρο για την πρόληψη και εμεί πιστεύουμε ότι η λύση του προβλήματος για την αντιμετώπιση της ρίζος παστικοποίησης είναι η πρόληψη. Σε λίγες μόνο εβδομάδες θα καταθέσουμε μια ειδική ανακοίνωση για τη ρίζος παστικοποίηση για να επεκτείνουμε λιγάκι την ανακοίνωσή μας. Όσον αφορά τώρα στο διαδίκτυο. Αναμφισβήτητα, ε, αυτό είναι προτεραιότητά μας. Εγώ προσωπικά μάλιστα συμμετέχω στις σχετικές συζητήσεις και μπορώ να σας πω ότι αυτή η πρόταση για μια κοινή πλατφόρμα αναφοράς για να μπορούμε να αποφύγουμε το εξής, δηλαδή ε, κάτι που παίρνει κανείς από μια πλατφόρμα να μπορεί να το μεταφέρει πολύ εύκολα σε μια άλλη πλατφόρμα και αυτό να επαναλαμβάνεται. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα, ενδιαφέρονται γι' αυτό, θα είναι μια συνεργασία ανάμεσα στις δύο ενδιαφερόμενες πλευρές και υπάρχει και ήδη ένα παράδειγμα, το Internet Forward Foundation είναι δηλαδή ε, ένας φορέας ιδιωτικού δικαίου και νομίζω ότι ο ιδιωτικός τομέας ενδιαφέρεται πολύ να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Κατά τα άλλα, έχουμε πει ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε κοινικοί, ε, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί την ευκαιρία ότι εδώ και καιρό υπάρχει απέτηση για μια νομοθετική πρόταση. Έχουμε επανειλημμένα διευκρινίσει ποιος είναι ο στόχος της πρωτοβουλίας. Σε ορισμένα κρατημέλη επικρατούν αυστηρότερες προϋποθέσεις ε, για προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεργαζόμαστε για να διευκρινίσουμε το κείμενο ε, στο πλαίσιο πάντα της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ γρήγορη πρόταση. Δεν ξέρω βέβαια, διερωτώ με τώρα πώς θα τα εφαρμόσετε όλα αυτά στην πράξη. Μπρικίτε, μήπως θέλεις σύντομα να πεις κάτι. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί ενδέχεται να υπήρξε κάποια παρεξήγηση. Εγώ δεν ρώτησα το τι θα γίνει αφού θα έχουν εφαρμοστεί όλα τα μέτρα, ε, κατά πόσο ενδεχομένω θα χρειαστούν επιπρόσθετα μέτρα. Ήταν λίγο πολύ ρητορική η ερώτησή μου. Με την έννοια ότι εγώ ανησυχώ. Δηλαδή, αν τελικά εφαρμόσουμε τα πάντα και παρόλα αυτά προκύψουν και άλλες επιθέσεις, τότε Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε τι είδους επιπρόσθετα μέτρα θα μπορούσαμε να λάβουμε ε, στο επίπεδο του ελέγχου και της αστυνομικής παρακολούθησης. Και κάνω αυτή τη ρητορική ερώτηση γιατί είμαι πεπισμένη ότι παρότι βέβαια πρέπει να ελέγξουμε την πολιτική μας της ασφάλειας, μόνο εφόσον εστιάσουμε στην παρακολούθηση και στα περιοριστικά μέτρα, αυτό μόνο δεν σταματάει την, την τρομοκρατία. Σας λέω, ήταν έτσι μια ρητορική ερώτηση για να στοχεύσουμε λιγάκι και σε άλλα θέματα και όχι μόνο ε, στην ασφάλεια. Ευχαριστούμε την Μπρικίτη και τα κράτη-μέλη που ε, συνέβαλαν σε αυτή τη συζήτηση και είμαι σίγουρος ότι κάποια από τα μέλη, κάποιοι από τους συνεργάτες μας ε, τη διάβασα την ανακοίνωση. δεν είναι πια και τόσο μακροσκελής, είναι επί της ουσίας και τίθεται το ερώτημα τι ακριβώς ε, πρέπει να κάνουμε, τι υπολείπεται στην εφαρμογή και ε, ειλικρινά θα τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρουσίασή σας και ευχαριστούμε και τα κράτη-μέλη που βρήκαν χρόνο να παρακολουθήσουν την συζήτηση. Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Συνάδελφοι, τώρα λοιπόν πάμε Νομίζω η Μαρία έχει ήδη έρθει και περιμένει υπομονετικά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λιγάκι νωρίτερα αν δεν διαφωνούν οι συνάδελφοι. Υποτίθεται θα ξεκινάγαμε στις 5, αλλά αν συμφωνούν και οι συνάδελφοι να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Πρόκειται για το σχέδιο συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για βραχία διαμονή. Θα μπορούσα ίσω να προβώ σε μια μακρά εξήγηση του θέματος, αλλά καλύτερα Μαρία, κυρία Γκαμπριέλ, να το κάνετε εσείς αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω ορισμένα πράγματα. Ως αποτέλεσμα της ε, τροπολογίας 53-29 του 2001 το Περού είναι μία από τις χώρες που θα περάσει από το παράρτημα 1 στο παράρτημα 2. Εκεί είναι οι τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται τις υποχρεώσεις θεώρησης όταν ε, περνάνε από τα σύνορα μιας τρίτης χώρας. Επίσης, ε, εμείς είμαστε μία από τις λίγες χώρες που ε, περάσαμε αυτόν τον έλεγχο πριν η Κομισιόν ε, αναλάβει την υποχρέωση να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για βραχία διαμονή για το Περού. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω του ότι έχει υπάρξει εδώ μεταξύ πολύ μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την ασφάλεια και την οικονομική κατάσταση στο Περού, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν επιπρόσθετοι λόγοι για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους κατοίκους του Περού. Το 2015 μονογράψαμε τη συμφωνία για αυτή την απαλλαγή η οποία τέτοια ισχύει 16 Μαρτίου του 2016. Κάθε φορά που συζητάμε τις θεωρήσεις θέλω να σας επισημάνω ότι οι συμφωνίες για απαλλαγή θεώρησης για βραχία διαμονή, αυτό πάντα είναι μία βελτίωση και σίγουρα αφορά το Περού. Επίσης, είναι μία ε, βελτίωση προς την κατεύθυνση των πιο στενών οικονομικών και πολιτικών σχέσεων. Αναβαθμίζεται ο πολιτικός διάλογος συμπεριλαμβανομένων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Εξάλλου, αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει στη βελτίωση της περιφερειακής συνοχής το Περού είναι μία από τις λίγες χώρες στη Λατινική Αμερική ε, του οποίου οι υπήκοοι πρέπει να έχουν θεώρηση να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτή η συμφωνία θα βοηθήσει και τις εμπορικές σχέσεις, ε, θα βοηθήσει τις επενδύσεις. Να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Περού, ε, σημαντικός στόχος για τις εξαγωγές μας. Η άρση λοιπόν της ε, θεώρησης θα διευκολύνει τις επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στο Περού. Όσον αφορά τώρα τους δρόμους που θα ανοίξουν με αυτή τη συμφωνία για να υπάρχει έτσι ένας ερωτημένος, βελτιωμένος πολιτικός διάλογος, θεωρώ ότι και αυτό θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ως προς την κινητικότητα, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεχής βελτίωση της συνεργασίας με το Περού για θέματα μετανάστευσης. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ε, σχετικά με το ποσοστό των ε, θεωρήσεων που απορρίφθηκαν. 6,1% το 2014 και 3% το 2015. Όμως να μην ξεχνάμε ότι Πρόκειται για διαβατήρια με βιομετρικά δεδομένα. 31 Δεκεμβρίου του 2015 ήταν ε, η αρχή εφαρμογής αυτού του νέου καθεστώτος. Ε, στο Περού υπήρχαν κάποιες δυσκολίες να εισάγουμε τέτοιου είδους ε, διαβατήρια και εμείς τα εισαγάγαμε τελικά μετά το Φεβρουάριο αντί για Ιανουάριο. Συγχαίρω λοιπόν την κυβέρνηση του Περού για την εκστρατεία ενημέρωσης για να προβληθούν τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας με τις θεωρήσεις ε, και το θέμα της μετανάστευσης. Να σας πω για άλλη μια φορά ότι το Περού έχει τη δυνατότητα να γίνει σημαντικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Θα θυμάστε όταν μιλάγαμε για την Κολομβία ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν η στρατηγική συμφωνία με τη Europol, μια συμφωνία που είχε υπογράψει το Περού. Το Περού ήταν ιδιαίτερα πρότιμο να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία με τη Europol και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τελειώνοντας λοιπόν θα αναφέρω άλλα δύο θέματα. Το ένα αφορά στην εγγύηση της δίκαιης αμοιβαιότητας. Ε, αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τα παρακολουθεί όλα εκ του σύναγκες και εμείς έχουμε αναλάβει από την πλευρά μας ιδιαίτερες ε, Ευθύνε και υποχρεώσει. Δεύτερον, αυτή η συμφωνία για τις θεωρήσεις ε, θα προβλέψει και μία μεταβατική περίοδο πριν από την επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προφανώ και στη διαδικασία αυτή πρέπει να είναι εταίρος επίσης όρης και θέλουμε να ελπίζουμε ότι το Περού θα είναι η τελευταία περίπτωση ε, όπου υπογράφεται μια συμφωνία με μια χώρα πριν εκφράσει το Κοινοβούλιο την άποψή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους και οδησηγητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είχαμε επικοδομητική, τακτική ανταλλαγή απόψεων και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η διορία είναι 3 Μαΐου για την κατάθεση τροπολογιών. Και στο πλαίσιο της διαδικασίας θα υποβληθούν μόνο τροπολογίες επί της διαδικασίας. Υπάρχει κάποιος ε, που θέλει να μιλήσει που είναι εδώ και περίμενε και πολύ ώρα να μιλήσει. Στρέφομαι όμως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ ολοκληρωμένη έκθεση για τους κινδύνους της παράτυπης μετανάστευσης, για τα βιομετρικά διαβατήρια, για την Europol. Όλα έχουν καλυφθεί μέσα στην έκθεση. Στις 17 Μαρτίου εδώ Ήδη παρουσίασα τη συμφωνία παρέκκληση από τη θεώρηση για το Περού, μια συμφωνία πρότυπο που συνάδει πλήρως με αυτό που συνηθίζουμε, περιλαμβάνει πολλά χρήσιμα στοιχεία, υπάρχει κοινή δήλωση στη συμφωνία όπου παρουσιάζονται οι όροι για την αναστολή της εφαρμογής της, εάν δεν τηρούνται το προαπαιτούμενα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνεργασία, τις επανειστοχέ και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, το έχω ήδη παρουσιάσει στην Επιτροπή σα. Να μιλήσω για την αμοιβαιότητα, Επομένω, δεν χρειάζεται θεώρηση για να πάνε στο Περού οι Ευρωπαίοι πολίτε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να πω σήμερα. Αν έχετε ρωτήσει στη διάθεσή σα, Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κυρία Γκαμπριέλ, θέλετε να επανέλθετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα να υποβάλω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας δίνετε ένα χρονοδιάγραμμα, μπορείτε. Πότε θα εγκρίνει αυτά τα διαβατήρια το Περού. Αρκετές χιλιάδες εκδόθηκαν στις αρχές της χρονιάς. Τώρα όμως πώς έχει η κατάσταση. Ο Πρόεδρος, παρακαλώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απάντηση. Το Περού έχει ήδη εκδώσει βιομετρικά διαβατήρια, το ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2016 και δεσμεύεται να το οριστοκοποιήσει μέχρι τον Ιούλιο αυτής της χρονιάς. Από ό,τι έχω καταλάβει, από τις 7 Ιουλίου του 2016 και μετά, μόνο βιομετρικά διαβατήρια θα εκδίδονται και τα παλιά σταδιακά θα εξαλειφθούν και θα αποσυρθούν. Τώρα, όπως είχα πει και την πρώτη φορά που πήρα το λόγο εδώ, ε, αυτή δεν θα είναι η τελευταία συμφωνία που ε, παρουσιάζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της ε, τροποποίησης των διαφόρων καταλόγων. Ο Γενικός Διευθυντής έχει συντάξει επιτροπή και την, επιστολή και την έχει απευθύνει στην Επιτροπή σας και ανακοινώνει τέσσερις τελικές συμφωνίες που θα σας υποβάλλουμε λίγαν συντόμως που έχουν ήδη υπογραφεί. Για τη Μικρονησία, τα νησιά Μάρσαλ, τα νησιά Σόλομον και το Του Βαλού. Αυτές οι συμφωνίες λοιπόν θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης Λίαν, συντόμως και μπορούμε να τις συζητήσουμε. Να συζητήσουμε όλο αυτό το θέμα με αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Κύριε Πάλμαν, ευχαριστούμε και την κυρία Καπριέλ. Ευχαριστούμε όλους. Ολοκληρώνεται η εξέταση αυτού του ζητήματος. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η κυρία Βαλέρο δεν είναι εδώ. Όμως για το μέθο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι πάλι η συγγήτρια η κυρία Γκαμπριέλ. Όμως δυστυχώς δεν θα έχουμε διερμηνία ε, από τα Γεωργιανά ε, πριν τις 5 και 4. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα διακόψουμε για 10 λεπτά Πέντε και πέντε να ξαναξεκινήσουμε αν συμφωνείτε. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Διακόπτουμε μέχρι τις 5 και 5. Συνάδελφε, ε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα στους συναδέλφους που μόλις μπήκαν στην αίθουσα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε προχωρήσει πολύ γρήγορα. Δεν θέλω να το μαθαίνουν και οι άλλες επιτροπές. Ασυνήθιστο γι' αυτό, για μας. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είστε έτοιμοι συνάδελφε, για το θέμα που σας αφορά. Ναι. Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σε σχέση με την απαλλαγή θεώρησης βραχίας διαμονής για κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων από την Κίνα. Είστε η παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Αυτό είναι ένα θέμα ε, που ζητήθηκε η συνένεσή μας. Πρόκειται λοιπόν για το διπλωματικό διαβατήριο, αλλά πρόκειται επίσης ε, και για την άδεια όπως είμαστε εμείς ε, ανθρώπων να μπορούν να έρχονται στις Βρυξέλλες. Δεν νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή το να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις ε, πολιτικές ομάδες θα πρέπει να υπάρξει διάλογος ε, για τα προβλήματα που μπορούν να προκληθούν στις διάφορες πολιτικές ε, ομάδες. Υπάρχει θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παρεμφερή θέματα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε από αυτού. Εμείς θα καταθέσουμε μια, ε, ένα σχέδιο έκθεσης που θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο και κατόπιν τον Ιούλιο θα πρέπει να έχουμε καταθέσει τις τροπολογίες και μετά ε, θα περάσουμε στην ψηφοφορία το φθινόπωρο, από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα έχουμε δηλαδή αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε. Ακόμα δεν έχω ορίσει ακριβώς τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, αλλά θα επικοινωνήσω με τους σκιώτες βέβαια όταν καταλάβω και εγώ ποιοι είναι. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εξής. Μήπως μπορείτε να μας πείτε, έχετε έτσι μια εικόνα του πόσοι περίπου θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα. Έχετε δηλαδή συγκεκριμένα δεδομένα, αριθμούς. Νομίζω αυτό θα ήταν χρήσιμο να το γνωρίζει κανείς. Και κατόπιν έχω και μία ερώτηση που αφορά στους επισκέπτες Δεν ε, έχω ακόμα εξετάσει όλα τα έγγραφα. Μπας περιπτώσει, ίσως η Κομισιόν μπορεί να μας ενημερώσει λίγο καλύτερα. Αν το έκανε αυτό θα σας ήμασταν ευγνώμονες. Και αν μπορείτε και να μας ενημερώσετε και για τη συνεδρίαση της ε, Κοινή Επιτροπής για τη διαχείριση αυτής της συμφωνίας. Άρθρο υπαριθμών 7. Και από αυτού θα επιτιμούσα η Κομισιόν να μας δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω σε αυτή τη φάση. Ε, με ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ να ακούσω την άποψη της Επιτροπής. Ευχαριστούμε. Ε, για το γεγονό ότι ήρθατε λίγο πιο νωρί όπω είπε και συγγνώμη, σα πιέσαμε. Ε, για του κοιόδε τώρα, κύριε Αμπελόβα. Για του σοσιαλιστέ, ο κύριο Ντέλτον, για το ECR και κυρία Πεζιά για την ε, ΓΚΟΕ. Οπότε, δεν ξέρω αν σε αυτή τη φάση θέλετε να πάρετε το λόγο, κύριε Ντέλτον, για αυτό το θέμα. Δεν υποχρεώστε να το κάνετε. Ε, πρόεδρε, είναι επικίνδυνο να λέτε σε ένα πολιτικό ότι δεν χρειάζεται να μιλήσει. Ε, σε κάθε περίπτωση, πάντω, ε, εδώ το ζήτημα νομίζω πω δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση, είναι περισσότερο τυπική μορφή. Εκείνο που θα πρέπει να φροντίσουμε είναι να είμαστε θετικοί και εναρμονισμένοι σε ό,τι αφορά την προσέγγιση μα, τι σχέσει μα με την Κίνα. Οπότε, αναμένω με ενδιαφέρον τη συνεργασία μα με του υπόλοιπου αισιόδη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Ταλτών που ήσασταν τόσο σύντομο. Ε, τώρα μια σύντομη παρέμβαση να ακούσουμε από την Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, αλλά ε, επιτρέψτε μου εν συντομία να αναφερθώ λίγο στο γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε αυτή η ε, πρόταση σε σχέση με την Κίνα. Όπως γνωρίζετε, ε, η Επιτροπή διαθέτει έντολη για την, μια συμφωνία επανεισδοχής με την Κίνα από το 2000 και με συνέπεια έχουμε προσπαθήσει εδώ να φέρουμε στο διαπράγμα των διαπραγματεύσεων ε, την ε, Κίνα ε, για το ζήτημα των επανεισδοχών, αλλά μας είπε η Κίνα ότι δεν ενδιαφέρεται, μας το έχει πει επανελειμμένο, οπότε τα τελευταία δέκα χρόνια αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε σμάτιν να θυμάμαι την πόρτα της Κίνας σχέση με αυτό το ζήτημα. Ε, τώρα, σε συνέχεια του νέου συστήματος ε, πληροφοριών ε, θεωρήσεων, μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε μια νέα κατάσταση γιατί όλοι οι ετούντες θεώρηση θα πρέπει βέβαια να διαθέτουν και τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Αυτό βέβαια δεν άρεσε καθόλου στην Κίνα, ότι θα ήταν υποχρεωμένοι δηλαδή οι διπλωμάτες τους να δώσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα για να λάβουν μια θεώρηση εισόδου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο αποκτήσαμε, αν θέλετε, και έναν μοχλό για να στήσουμε περισσότερη πίεση στην ε, Κίνα. Οπότε στο πλαίσιο των διαλόγων ξεκίνησε μια συζήτηση και φτάσαμε σε μια συμφωνία πακέτο αν θέλετε, η οποία προβλέπει αφενό ε, την ε, συμφωνία από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για μια απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοση θεώρηση ε, για κατόχου διπλωματικών διαβατηρίων και από την πλευρά τη ε, Κίνα να επιτρέπει ε, στα κράτη-μέλη να ανοίξουν περισσότερα κέντρα επεξεργασία θεωρήσεων στην υπηρετική Κίνα. Και βέβαια ε, ε, μας επέτρεψε επίσης να ξεκινήσουμε ή ε, προβλέπει αυτή η συμφωνία πακέτο πρακτική έναρξη της συνεργασίας σε ό,τι αφορά τις επανεισδοχές. Αυτή ήταν η πρώτη αφορα τις αυτη ηταν η πρωτη φαση και τώρα στη δεύτερη φάση θα ξεκινήσουμε την διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας διευκόλυνσης του καθεστώς θεωρήσεων και μια πλήρη συμφωνία σε ό,τι αφορά τις επανεισδοχές. Αυτά λοιπόν είναι γενικότερου πλαισίου και επαφών για αυτό το ζήτημα γύρω από αυτό το ζήτημα και τώρα σε ό,τι αφορά αυτήν την ε, συγκεκριμένη συμφωνία είναι τυποποιημένη, δηλαδή ε, εξαίρεση σε ό,τι αφορά μόνο κατόχους διπλωματικών διαπατηρίων, αλλά για πρώτη ε, φορά έχουμε εφαρμόσει και αυτούς τους κανόνες λεσέ πασέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα βέβαια το οποίο τα αποδεί και προς όφελος και εδώ συναδέλφων από το Κοινοβούλιο. Κατά τα λοιπά προβλέπονται εδώ συγκεκριμένες διαδικασίες που θα εφαρμόζονται, ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα ωφεληθούν από αυτές τις διατάξεις και από εκεί και μετά, όπως αναφέρθηκε ήδη, ε, προβλέπει και την ε, δημιουργία μιας κοινή επιτροπής. Μια τέτοια κοινή επιτροπή αποτελεί μια, ένα πολύ τυποποιημένο στοιχείο τέτοιων ε, δηλαδή συμφωνιών διευκόλυνση του καθεστώτος θεωρήσεων ή απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοση θεώρηση. Όπως Όπω προβλέπει και το σχετικό άρθρο, αυτή η μεικτή επιτροπή έχει το καθήκον παρακολούθηση τη εφαρμογή τη συμφωνία. Αν υπάρξει οποιοδήποτε ε, ζήτημα σε επίπεδο εφαρμογή, για παράδειγμα καταχρηστική εφαρμογή ή ε, λαθρομετανάστευση ή ε, παραβίαση του χρόνου παραμονή με βάση τη θεώρηση, όλα λοιπόν αυτά τα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν μπορούν να συζητηθούν στο πλαίσιο αυτή τη κοινή επιτροπή προτού αποφασιστεί η λήψη σοβαρότερων μέτρων. επιτροπη προτου αποφαστει η ληψη σοβαροτερων μετρων τωρα σε ό,τι αφορά το ερώτημα που τέθηκε για ε, τα άτομα τα οποία μιλάμε, χοντρικά να σας πω, λιγότερα από 20.000 άτομα ως κατόχους δηλαδή διπλωματικών διαπατηρίων. Βέβαια στην ε, ε, πράξη θα έχουμε, ή μάλλον από την πλευρά μας έχουμε πολύ περισσότερους, έχουμε γύρω στα 100.000 άτομα τα οποία είναι κάτοχοι διπλωματικών διαπατηρίων, αλλά έχουμε τους και εκείνου που αποφελούνται από την ΕΣΥΠΑΣΗ, οι οποίοι βέβαια δεν είναι διάφορε χιλιάδε, αλλά λιγότερο. Ευχαριστούμε ε, τον ε, ΣΥΤΗ, τον κύριο Ντάλτον, ε, την ΣΥΤΗ, τον κύριο Ντάλτον και την Επιτροπή. Περνάμε τώρα στο σημείο 7 τη ημέρα τη διάταξη το γεγονός ε, δηλαδή ότι η κατοχή τρίτων ε, χωρών ε, θα πρέπει να είναι κάτοχοι θεώρηση, σχετική συμφωνία που προβλέπει την απαλλαγή από τη σχετική υποχρέωση και το ενδεχόμενο περίληψη και τη γεωργία σε αυτή τη συμφωνία. Θα ακούσουμε εδώ μία παρουσίαση από την πλευρά τη Επιτροπή. Για να κάνω μία, ή μάλλον πριν από την εισαγωγή, να πω ότι έχουμε στο κανάλι 25 την διερμηνία στα Γεωργιανά μάλλον το γνωρίζετε, αλλά όσο δεν το γνωρίζετε, στο κανάλι λοιπόν 25 για τα Ε, σε αυτό λοιπόν το τελικό, τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη έχουμε να κάνουμε με τον ε, κανονισμό του Συμβουλίου 539 ε, του 2001 ε, σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη της γεωργίας στην σχετική συμφωνία για την απαλλαγή της υποχρέωσης από την έκδοση θεώρησης μόνο με την, υπό την υποχρέωση της ε, συλλογής των ε, ε, βιομετρικών δεδομένων. Πριν από την έναρξη του σχετικού διαλόγου είχε συναυθεί μια συμφωνία διευκόλυνση έκδοση θεωρήσεων και μια συμφωνία επανεισδοχή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Γεωργία και οι δύο αυτέ συμφωνίε τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Μαρτίου του 2011. Η ε, Επιτροπή παρουσίασε στην γεωργιανή πλευρά ένα σχέδιο δράση για την απελευθέρωση του καθεστώτο θεωρήσεων ε, με βάση το οποίο παρακολουθήθηκε και η πρόοδο που έκανε η Γεωργία στο πλαίσιο τη για την εφαρμογή αυτή τη συμφωνία. Ε, στην δική μας ε, Επιτροπή έχουν γίνει σε παρουσιάσεις των εκθέσεων προόδου σε σχέση με αυτή τη συμφωνία και στην τέταρτη αυτή έκθεση προόδου που μας παρουσίασε η Επιτροπή θεώρησε ότι έχει, κάνει όλα, έχει εφαρμόσει όλα τα προαπαιτούμενα ε, για την εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας και με βάση αυτή την αξιολόγηση, με βάση την μου νομοθετική διαδικασία η Επιτροπή μας προτείνει τώρα αυτή την απόφαση. Οπότε ε, θα ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Ε, χαιρετίζω και καλωσορίζω εδώ και τα μέλη του ε, Γεωργιανού Κοινοβουλίου που βρίσκονται εδώ μαζί μα και τα, ε, και με του οποίου είχαμε συνεργαστεί και στο πλαίσιο και τη ε, δεύτερη ε, συνεδρία τη Βιομηχανική Συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργία. Και ε, καλωσορίζω εδώ και τον κύριο Σφιάρ Πατσαριντάτσε. Ε, ζητώ συγγνώμη για την κακή ε, προφορά. Ε, βέβαια γνωρίζω και τον κύριο Σεβαρντινάτσε και ζητώ συγγνώμη που πέρδεψα το όνομα ε, σας. Ε, βάση περιπτώσει. Σας καλωσορίζω θερμά. Ε, ε, δύο λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι, του κύριου Εκανή και ο κύριο Πατσαρτινάτσε είναι συμπρόεδροι. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στην Επιτροπή και μετά στην συγκεκριμένη και στον κύριο Καπρίλ και στους υπόλοιπους που θέλουν να πάρουν το λόγο και οποιοδήποτε άλλο βέβαια από τα μέλη της Επιτροπής που θέλει να πάρει το λόγο. Ε, να δώσω λοιπόν το λόγο καταρχήν στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Θα είναι επισύντομη η παρουσίασή μου, όπως, ε, γιατί ο Πρόεδρος συνόψισε το ιστορικό θα θυμάστε τις συζητήσεις στην Επιτροπή σας για, την, για το σχέδιο δράσης απελευθέρωσης από την υποχρέωση θεώρησης. Στις 18 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την τέταρτη και τελευταία έκθεση προόδου για αυτό το σχέδιο δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπέρανε ότι... Ε, όλοι οι στόχοι είχαν εκπληρωθεί και επομένως στις αρχές του 2016 θα παρουσίαζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της. Τον Ιανουάριο έγιναν διάφοροι γύροι συζητήσεων στο Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη επιβεβαίωσαν την αξιολόγηση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Γεωργία πλήρει όλες τις ε, προϋποθέσεις που προβλέπει το σχέδιο δράσης απελευθέρωσης της θεώρησης και αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα και κατάληξη των συζητήσεων στο Συμβούλιο. Συνεπώς, στις 9 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε την πρότασή της, η οποία είναι απλή. Ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιηθούν τα παρατήματα του κανονισμού 539 που είναι ο σχετικός κανονισμός για τις θεωρήσεις και η γεωργία να μεταφερθεί από το παράρτημα 1 στο παράρτημα 2. Το πρώτο είναι ο, ο κατάλογος των χωρών τον οποίο οι πολίτες πρέπει να φέρουν θεώρηση και παράρτημα 2 είναι οι χώρες που οι πολίτες τους δεν χρειάζεται να φέρουν θεώρηση βίζα για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Διευκρινίζεται βεβαίως ότι αυτό ισχύει για τους κατόχους των βιομετρικών, διαβατηρίων που είναι ε, εκδοθέντα βάσει των διεθνών προτύπων. Επομένως ε, θα συνεχίσει να ισχύει η υποχρέωση θεώρησης για όσους δεν έχουν βιομετρικά διαβατήρια γεωργιανούς και θα υπάρξουν εκεί οι συμφωνίες διευκόλυσης για τις θεωρήσεις. Θα συνεχίσουν να ισχύουν αυτές οι συμφωνίες. Τώρα για την πρόταση αυτή καθεαυτή η Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι η παρέκκληση από τη θεώρηση δεν χρειάζεται να είναι αντικείμενο ξεχωριστής συμφωνίας. Θα είναι άμεσα εφαρμοστέα η απόφαση 20 μέρες μετά την δημοσίευση του τροποποιηθέντος κανονισμού στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αυτό που ενδιαφέρει τα μέλη της Επιτροπής σας είναι ότι ένα έγγραφο εργασία σε τεχνικό επίπεδο έχει προσαρτηθεί στην τέταρτη έκθεση προόδου και γίνεται αξιολόγηση για τις μεταναστευτικές ροές, για τον αντίκτυπο στην ασφάλεια, ενδεχομένω σας ενδιαφέρει να το διαβάσετε, γιατί σχετίζεται με την πρόταση και τέλος στο επεξηγηματικό υπόμνημα της πρότασης θα βρείτε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχίσει να παρακολουθεί το πώς η Γεωργική εφαρμόζει αυτά τα προαπαιτούμενα μέσα, μέσα από τις υφιστάμενες δομές και, εάν χρειαστεί, μέσα από μηχανισμούς ad hoc επιτόπου. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Με χαρά δίνω το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια κυρία Καμπριέλ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Γεωργίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρέμβασή της. Ως εισηγήτρια για το θέμα αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξή μου στην νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την παρέκκληση από την υποχρέωση θεώρησης για τους γεωργιανούς κατόχους βιομετρικών διαβατηρίων όταν αυτοί ταξιδεύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή που η νομοθετική αυτή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε βάση αξιολόγηση στην τέταρτη και τελευταία έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή από πλευρά γεωργίας του σχεδίου δράσης για την απελευθέρωση από τη θεώρηση φαίνεται ότι η Γεωργία έχει κάνει την απαραίτητη πρόοδο και έχει προβλέψει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να εγγυηθεί την ε, ε, βιώσιμη εφαρμογή όλων των κριτηρίων, δηλαδή την εφαρμογή όλων των κριτηρίων σε βάθος χρόνου, επιμονή μου βάσεως. Και άρα Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει τους γεωργιονούς πολίτες και θα συσφίξει τις οικονομικές και πολιτισμικές μας σχέσεις. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Εκτιμούμε ιδιαίτερο τις οργανωτικές προσπάθειες που έχει καταβάλει η Γεωργία στο δεύτερο εξάμεινο του 2015 και μάλιστα προόδευσε η χώρα αυτή και σε τομείς και σε παιδεία που είχαν καχεκτική πρόοδο στο παρελθόν. Έγιναν μεταρρυθμίσεις πολύ σημαντικές σε θέματα μετανάστευσης, σε θέματα πολιτικής ασύλου, διαφθοράς, ε, νομιμοποίησης παράνομων προσόδων, σε θέματα καταπολέμησης όλων αυτών, καταπολέμησης των ναρκωτικών και άλλων σοβαρών ε, αδικημάτων, ποινικών αδικημάτων. Πρέπει λοιπόν να στείλουμε αυτό το θετικό μήνυμα γιατί η Γεωργία έχει παρετηθεί του δικαιώματος να ζητά θεωρήσεις για Ευρωπαίους πολίτες που θα μείνουν στη Γεωργία μέχρι 90 μέρες. Και επειδή ε, είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολόθερμα υπέρ της αμοιβαιότητας και επειδή έχουν υπάρξει όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις από πλευράς Γεωργίας, εμείς στηρίζουμε την πρόταση αυτή. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες και έχω δύο ερωτήσεις να θέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, Ποιο είναι το ποσοστό των ετοιμάτων για θεώρηση που την χάνουν απόρριψης και ποια είναι η κυρία αιτιολογία για την απόρριψη. Ξέρουμε ότι το ποσοστό των θεωρήσεων που, έχει, που έχουν απορριφθεί πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με ένα ομοιόμορφο αναλυτικό σύστημα μετανάστευσης. Αυτό σημαίνει ότι θα συγκεντρώνονται στοιχεία από όλες τις κρατικές υποδομές για τη μετανάστευση ε, προς τη χώρα ή από τη χώρα. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό για να έχουμε σαφή εικόνα ε, της ανάλυσης κινδύνου θέματα που μπορούν να γίνουν αντικείμενο καλύτερης διαχείρισης μέσα από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τέταρτη έκθεση προόδου της Επιτροπής λέει ότι πρέπει να δοκιμαστεί το σύστημα μέχρι τα μέσα του 2016. Έχετε πληροφορίες ε, πόσο έχει προχωρήσει η Γεωργία στο θέμα αυτό. Ε, Αυτά είναι θεμελιώδη ζητήματα για εμένα και θα ήθελα να τα τονίσω σε αυτό το στάδιο. Πρέπει τις προκλήσεις να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες. Άλλωστε, όταν συζητείτε μια ε, τέτοια έκθεση, είναι πολύ σημαντικό να είναι ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχουν εκπρόσωποι στις Επιτροπές Παρακολούθησης. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετέχουν στις συζητήσεις. Και θέλω να ξαναπώ το εξής. Κάθε φορά που συζητούμε για τις θεωρήσεις, το μόνο που πρέπει να είναι στο μυαλό μας, να βρίσκεται στο μυαλό μας, είναι οι πολίτες. Αυτά υπάρχουν για, και είναι προς όφελος των πολιτών. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη και να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες για την ανάληψη θετικής δράσεις και αυτά θα βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ Γεωργίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσει η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα κύριε Καρίμ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα το ότι ε, μπορώ να προεδρεύω στην Επιτροπή σας. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω, να καλωσορίσω εδώ τη Γεωργιανή ε, Αντιπροσωπεία. Ε, καλωσορίζω και τον φίλο μου και τα μέλη του Κοινοβουλίου και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, περιλαμβανομένου και του Υπουργού Δικαιοσύνη που είναι παρόν στην αίθουσα. Θα ήθελα επίση ε, να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μου την κυρία Γκαμπριέλ για όλα αυτά που μας είπε η προσέγγιση που έχει υιοθετήσει κατά την άποψή μου είναι μια πολύ καλή προσέγγιση για το κοινοβούλιο μας. Και Συγχαίρω επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Ε, έχουν καταστήσει απόλυτα σαφές ότι σε κάθε ευκαιρία που τους δόθηκε ε, να έρθουν σε επαφή με τη γεωργιανή πλευρά. Ε, η γεωργιανή πλευρά τα καταφέρε μια χαρά μετά από μια μακρά διαδικασία και έτσι λοιπόν η Επιτροπή μας και ο εισηγητής νομίζω ότι θα έχουν τελικά την εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη και όλα αυτά να βασίζονται στην ευρύτερη προσέγγιση που έχουμε επιτήσει ευθύς εξ αρχής. Η προσέγγιση μας δηλαδή ήταν να περάσουμε ένα μήνυμα, το μήνυμα της αλληλεγγύης με τους πολίτες της Γεωργίας. Η συνάδελφός μου πολύ σωστά λέει ότι εδώ διακυβεύεται το μέλλον των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε την προσέγγιση της γεωργίας έναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση ε, εκπέμπει λάθος μήνυμα και κυρίως ε, σε τομείς όπως είναι η Νότια Οσετία γιατί εκεί τα μηνύματα μπορούν να ερμηνευτούν πολύ αρνητικά και το θέμα είναι ότι πρέπει να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη στο σύνολο της ε, εδαφικής ακερότητας και της ε, κυριαρχίας της Γεωργίας. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές προσεγγίσεις από το πώς, ε, πάρα πολλές επιπτώσεις από το πώς θα προσεγγίσουμε το θέμα. Σύμφωνα με αυτά που είπε η κυρία Γκαμπριέλ, ε, τα στηρίζω, ελπίζω ότι και εκείνη θα στηρίξει τη δική μου την πρόταση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που προτείνω. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε και εσάς ε, και Τώρα ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Συμπρόεδρο της Επιτροπής Σύνδεσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος γιατί εδώ βρισκόμαστε στην αίθουσα της Άννα Λίντ και πρέπει να σας πω ότι ήμουν πανευτυχής νιώθω πανευτυχής γιατί είχα την χαρά και την τιμή να τη γνωρίζω προσωπικά και ακόμα και τώρα θυμάμαι τις συναισθηματικά φορτισμένες συζητήσεις μας για το μέλλον της Γεωργίας, για τον δρόμο που θα ακολουθούσε η Γεωργία το 2001 τότε όταν ήμουν στο ε, Υπουργείο Εξωτερικών, ε, στο Μπακού και η κυρία Λίντε ήρθε ως εκπρόσωπος μιας ε, τρόικα εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μπακού. Έχετε απόλυτα δίκιο κυρία Γκαμπριέλο ότι πρόκειται για τους Γεωργιανούς, για τους πολίτες Ρίχνοντας λοιπόν μια ματιά στην ιστορία, διαπιστώνουμε ότι η Γεωργία με την παράδοση που έχει, με τον πολιτισμό της και τις φιλοδοξίες της, ανέκαθεν ήταν μέλος της Ευρώπης. Η Γεωργία ε, θεωρούσε ότι η ανάπτυξη την οδηγεί ε, μόνο μέσα στην Ευρώπη. Επίσης ε, η Γεωργία ανέκαθεν αναγνώριζε ότι ο μόνος τρόπος για να υπερασπιστεί τους πολίτες της είναι η ε, προσήλωση στις ευρωπαϊκές αξίες. Πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι για τη Γεωργία η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σταθερότητα, η δημοκρατία, η ισότητα και η ευημερία. Ο στόχος, ο δρόμος για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι να παραμείνει κανείς συνδεμένος με την ε, ευρωπαϊκή κοινωνία, ε, την επιστήμη, αυτή η έννοια της ε, ευρωπαϊκής κοινωνίας εξακολουθεί να υπάρχει, αναβιωμένη μάλιστα σήμερα. Βλέπουμε ότι ό,τι θέλουμε να πετύχουμε για το μέλλον έχει ρίζες στο παρελθόν. Οι πρόγονοί μας κατάλαβαν ότι η χώρα μας μπορεί να είναι ζωντανή μόνο μέσα από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών αξιών. Εμείς λοιπόν οι Γεωργιανοί βρισκόμαστε στην πόρτα της ευρωπαϊκής οικογένειας και έχουμε την τιμή να σας ανακοινώσουμε ότι θέλουμε και εμείς να ενταχθούμε σε αυτήν την κοινωνία που ανήκουμε ιστορικά. Η κυβέρνησή μας προσπαθεί να μας φέρει πιο κοντά στο στόχο αυτό και σήμερα Έχουμε την ε, χαρά να βιώνουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τις ε, προσπάθειές μας. Ε, θέλουμε να μπορούμε να προσβλέπουμε στη δική σας την υποστήριξη και την υποστήριξη των Ευρωπαίων συναντέλφων σας. Πολλοί συμπατριώτες μας στη Γεωργία πολίτες της Γεωργίας, η Απχαζία και η Νότια Σετία προφανώς και ανήκουν στη δική μας τη χώρα, αυτοί όλοι παρακολουθούν αυτή τη συνεδρίαση και ελπίζουν να μπορέσουμε και εμείς να ενταχθούμε σε αυτήν την οικογένεια όπου ανέκατεν ανήκαμε. Σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε τη δυνατότητα να πούμε αυτά τα λίγα λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ για την αντιπροσωπεία σας, η οποία βρίσκεται εδώ μαζί μας. Ε, ναι, υπάρχει streaming και προφανώς οι φωνές ακούγονται και εκτός αυτής της αίθουσας. Νομίζω πως ε, ε, θα έπρεπε να δώσω το λόγο και πάλι στην κυρία εκτός και αν η Επιτροπή θέλει να κάνει μια σύντομη παρέμβαση. Καλώς. Η Επιτροπή λοιπόν για μια σύντομη παρέμβαση και μετά συγγήτρια. Ε, Πρόεδρε, ναι, πολύ σύντομα να απαντήσω σε δύο ερωτήματα που έθεσε εσύ. Το πρώτο αφορούσε τα δικαιώματα άρνηση ε, ε, θεώρηση στη Γεωργία και ε, να πούμε ότι στο τελευταίο, το τελευταίο το ποσοστό αυτό των αρνήσεων δηλαδή ήταν γύρω στο 12,5% παρότι εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανά κράτος μέλος. Ε, και μας ρωτήσατε επίσης σε ό,τι αφορά τους κυρίους λόγους για αυτή την άρνηση ε, και ποιες πληροφορίες έχουμε με βάση την, τον τοπικό φορέα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στο επίπεδο του χώρου Σέγγεν. Ε, οι κύριοι λοιπόν λόγοι για την άρνηση ήταν η παρουσία υποβολή ενός υποστηρικτικού εγγράφου το οποίο ήταν όμως δεν ήταν γνήσιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα που μου θέσατε και το οποίο αν δεν απατώμε έχει να κάνει με το σύστημα διαχείρισης μετανάστευση. θα ήθελα εδώ να δώσω το λόγο εδώ στον συναδελφό μου για να το απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ τον Πίας και ευχαριστούμε για αυτό το ερώτημα σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση της μετανάστευσης. Ένα-δύο σημεία που θα ήθελα να θίξω σε ό,τι αφορά ε, την ε, διαδικασία απελευθέρωσης του, της έκδοσης θεωρήσεων ή ο μηχανισμός διαχείρισης μετανάστευσης βελτιώνεται, έχει βελτιωθεί και έχει αξιολογηθεί από τους εμπειρογνώμονες των κατομελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οριστικοποιήθηκε το 2014 με μια νέα νομοθεσία σε ό,τι αφορά το νομικό καθεστώς ε, των αλλοδαπών και των απάτριδων και επίσης ε, το νομικό πλαίσιο άλλαξε και με την ε, ένα νέο τμήμα για τα ζητήματα μετανάστευσης, το οποίο αποτελεί πλέον τμήμα του Υπουργείου Στουρκών από το Δεκέμβριο του 2014 και μέσα στη δεύτερη φάση ε, του σχεδίου δράσης της ε, εφαρμογή του καθεστώτος απελευθέρωση και εδώ αναφέρουμε δηλαδή στην επιχειρησιακή πλευρά των ε, σχετικών μεταρρυθμίσεων να πούμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2015 δημιουργήθηκε ένα ε, πλήρε ε, σύστημα αξιολόγηση κινδύνων συμπληρωματικά προ το εφιστάμενο ε, νομικό πλαίσιο και έτσι χάρη σε αυτό το νέο σύστημα η συλλογή των δεδομένων για του σκοπού τη διαχείριση τη μετανάστευση θα λαμβάνει χώρα από την πλευρά 7 διαφορετικών υπηρεσιών τη Γεωργία και όχι μόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών όπω γίνονταν μέχρι τώρα. Νομίζω, ελπίζω να απάντησα στο ερώτημά σας, πάντως το σκεπτικό είναι να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει ε, ε, ε, σε επίπεδο μετανάστευση Γεωργίου, τόσο ώστε να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε και τις τάσεις οι οποίες μπορούν να αναδειχθούν. Ευχαριστούμε την Επιτροπή και κυρία Γκέμπρε λοιπόν, για να κλείσουμε το αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα να πω δύο λόγια. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις που μου έδωσε στα δύο ερωτήματα που έθεσα. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Καρίμ που συμμετείχε στις συζητήσεις και να διαβεβαιώσω τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ότι το μήνυμα του, τα μηνύματα των γεωργιανών πολιτών ε, τα ακούσαμε, ε, τα λάβαμε, η διαδικασία θα συνεχιστεί κανονικά ε, και θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους κοιόδες εισηγητές. Um, ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για μία ακόμα φορά για την παρουσίαση αυτή. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους, τους δύο εδώ και όλους τους εκπροσώπους από την της Γεωργίας και του Κοινωνικού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας σήμερα εδώ μαζί μας στην Επιτροπή ΛΕΜΠΕ. the next uh, ε, συνάδελφοι, τη ε, 13 ε, ...30 Απριλίου